Members, if you could take your seats. Members, if you could take your seats, please. Thank you very much. Um, I would... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη των Επιτροπών Γιούρη και Αύκο μαζί με τα μέλη της ε, Ήτρε και της ΑΦ... Ε, Πέτη που είναι συνδεδεμένα. Ευχαριστώ πολύ ε, που ήρθατε για την ακρόση και καλωσορίζω και τον υποψήφιο Επίτροπο Σεύσοβιτς για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις. Θα προεδρεύσει η Επίτροπη Γιώρη σύμφωνα με τον κανονισμό το παράρτημα 7 και θα εξετάσουμε την ευρωπαϊκή του προσήλωση, την προσωπική του ανεξαρτησία, ε, καθώς επίσης και τη γνώση ε, του χαρτοφυλακίου και τις ικανότητε επικοινωνίας. Ε, θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο απευθείας και θα υπάρξει και βίντεο. Θα θυμάστε ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αφού εξέτασε τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του υποψηφίου αντιπροέδρου, δεν εξέφρασε αντιδράσεις για τη διεξαγωγή ε, της ακρόασης. Ε, ενημερώνω ότι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος θα κληθεί να κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση μέχρι ένα τέταρτο. Στη συνέχεια, 25 ερωτήσεις θα τεθούν ε, ανά ε, μία ερώτηση από ένα μέλος ε, ενός λεπτού και δύο ε, λεπτά απάντηση από τον Αντιπρόεδρο υποψήφιο με τη δυνατότητα το ίδιο μέλος να κάνει υπερώτηση ενός λεπτού με μονόλεπτη απάντηση από τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο. Καλησπέρα σε όλους. Να θυμίσω στα μέλη των Επιτροπών Αύκο και Γιούρι ότι σας έχει επιδοθεί το βιογραφικό σημείωμα του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς και επίσης σας έχουν δοθεί οι γραπτές απαντήσεις, τις γραπτές ερωτήσεις που του είχατε υποβάλει. Να θυμίσω επίσης στον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς που δεν είναι για πρώτη φορά βέβαια ενώπιον του ε, Κοινοβουλίου αλλά για τρίτη μάλιστα φορά ως Επίτροπος ότι δηλαδή η ακρόασή μας θα διαρκέσει μέχρι τις 17.30. Ένα τρίωρο δηλαδή. Είμαι πολύ ικανοποιημένο ως πρόεδρος της ΑΦΚΟ αλλά και ως πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το χαρτοφυλάκιο του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς περιλαμβάνει την συνέχεια που σκοπεύει να δώσει η Επιτροπή στα αιτήματα ε, ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει ξεκινήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια δέσμευση, κύριε Αντιπρόεδρε, που επισήμως σας ζητώ εσείς έχετε διατελέσει επίτροπος στην Επιτροπή ε, Μπαρόζο και έχετε ήδη υπάρξει υπεύθυνο για τις σχέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο μάλιστα με πολύ ε, ε, καλή, καλές επιδόσεις, αλλά όμως δεν θέλουμε να σας ζητήσουμε να δεσμευτείτε μόνο τύπης, για να έχει το Ευρωκοινοβούλιο πλήρη εξουσία. Δηλαδή να είναι ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο να έχει το δικαίωμα νομοθετική πρωτοβουλία. Βεβαίω έτσι να μπορεί να μετατρέψει σε συγκεκριμένε ενέργειε, ε, τι δεσμεύσει που ανέλαβε η ε, πρόεδρο Φοντερ Λόιεν αλλά και εσεί, ο ίδιο. Για μα αυτό είναι προτεραιότητα. Εάν θέλουμε να περιορίσουμε την απόσταση ανάμεσα στου πολίτε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να μένει ε, μόνο ο διεκπαιρεωτής. Βεβαίως, έχουμε δεσμευθεί ε, και έχετε δεσμευθεί και ε, για εξουσίες ερευνητικές για το Ευρωκοινοβούλιο. Για μας το, εδώ αποτελεί αυτό άλλη μια προτεραιότητα. Είμαι βέβαιος, πως, όπως έχετε κάνει και στο παρελθόν, όταν ε, είχατε αναλάβει τις διαθεσμικές ε, σχέσεις θα ε, εργαστείτε ώστε να υπάρχει μια πραγματική ανάμεξη και εξουσία στο Κοινοβούλιο, δηλαδή να περιοριστεί έτσι η απόσταση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες, αλλά και η απόσταση ε, ε, και οι θετικές σχέσεις ανάμεσα σε Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο να μπορέσουν να ε, ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο. Συνήθως ε, κάποιες προσπάθειες συνεργασίας μπορεί να σκοντάψουν σε υπερβολικό γραφειοκρατικό ε, φόρτο, αλλά θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι θεσμοί, ε, Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο να μπορέσουν να συνεργαστούν αγαστά και ομαλά. Θα ήθελα επίσης να πω στον ε, Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς αλλά και σε όλους τους συναδέλφους ότι αντίθετα με αυτό που έκανα όσο ήμουν πρόεδρος, δηλαδή ήμουν πολύ ευέλικτος όσον αφορά το χρόνο Σε τούτη εδώ την περίσταση δεν θα μπορέσω να είμαι τόσο ελαστικός, όπως ε, θύμισε η πρόεδρος Δετσίνκα. Έχετε ερωτήσεις για δύο λεπτά. Μπορείτε να κάνετε επερώτηση μέσα στο πεντάλεπτο και μετά έχουμε τη σύντομη απάντηση του Επιτρόπου σε ε, το face to face. Λοιπόν, θα ξεκινήσει αμέσως μετά από την αρχική εισήγηση του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς, στον οποίο και δίνω αμέσως το λόγο για 15 λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε Νετσίνκα, αγαπητέ Πρόεδρε Ταγιάννη, αξιότιμοι αντιπρόεδροι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Όντως ε, με τιμά ιδιαιτέρως η παρουσία μου εδώ παρουσία μου εδώ ως υποψηφίου επιτρόπου και νιώθω μεγάλο προνόμιο που εγώ εγκαινιάζω αυτή την εβδομάδα συζητήσεων και ελέγχου που παρουσιάζουν την καλύτερη μορφή της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Φυσικά υπάρχει ένα συναισθηματικό στοιχείο σε αυτά, γιατί σε λίγες εβδομάδες θα εορτάσουμε τα 30 χρόνια ελευθερίας στην πατρίδα μου τη Σλοβακία, μετά τη Βελούδινη Επανάσταση. Και θυμάμαι πολύ καλά πώς κοιτούσα αυτό το διαβόητο παραπέτασμα μέσα από τα σιδηροπλέγματα, σιδηροφλάγματα και κοιτούσα το Δούναβι και δεν μπορούσα να φανταστώ εκείνη τη μέρα που θα μπορούσα να τον περάσω και να πάω στην Αυστρία να εργαστώ για μια ε, Ενωμένη Ευρώπη. Και η εμπειρία μου αυτή συνέβαλε στην ακράδαντη πεποίθησή μου ότι οφείλουμε να δημιουργήσουμε το μέλλον μας ως Δημοκρατικής Ένωσης και σέβομαι ιδιαίτερα τους κοινού μας θεσμούς και αξίες. Και αυτό είναι πολύ πιο προφανέ σήμερα που οι παγκόσμιες αλλαγέ έχουν ένα προηγούμενο ρυθμό. Το οικολογικό αποτύπωμα τη ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει μια πραγματικά επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. και η παγκόσμια κούρσα για την τεχνολογική προ... πρωτοκαθεδρία θα μεταμορφώσει τα οικονομικά μα μοντέλα και τι κοινωνίε μα. και σίγουρα η πολυμέρεια βρίσκεται υποποίηση και η εποχή τη παραπληροφόρηση μαζί με τις συνεχείς ανισότητες Δημιουργούμε μια δοκιμασία για τη δημοκρατία μας. Οπότε αντιμετωπίζουμε ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς θα εξασφαλίσουμε να μην καταλήξουμε μια μεσαία δύναμη εγκλωβισμένη ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Κίνα. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει, είμαι πεπισμένο ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 10 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η λειτουργία μα θα εδράζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Γι' αυτό πραγματικά με τιμά ιδιαίτερο το γεγονό ότι η εκλεγμένη ε, πρόεδρο. Ε, ε, με επιφόρτισε με το χαρτοφυλάκιο της, ε, των διοργανικών ε, σχέσεων και της πρόβλεψης. Και σίγουρα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φυσικοί εταίροι. Έχουμε θέσει στέρα θεμέλια της συνεργασίας μας και προτεραιότητά μου θα είναι να αναβαθμίσω αυτή τη συνεργασία σε μια ξεχωριστή εταιρική σχέση που θα βασίζεται στην μεταξύ μας εμπιστοσύνη αλλά και στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Γι' αυτό προτείνω η εταιρική μας σχέση να υπερβαίνει το νομοθετικό τομέα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια του πολιτικού κύκλου κατά την συγκέντρωση τεκμηρίωσης και την πρόβλεψη για να διαμορφώσουμε από κοινού την πορεία της Ευρώπης. Κοινέ προτεραιότητες και κοινό πρόγραμμα εργασιών και ένα νέο δικαίωμα πρωτοβουλίας που είναι πολύ σημαντικό για σας, καθώς και καλύτερη εφαρμογή με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ε, τρόπο διαχείριση των κρίσεων με ω επιτοπλίστων διακυβερνητική προσέγγιση. Ένα ισχυρότερο κοινοβούλιο χρειάζεται και μια ισχυρότερη και πιο νομιμοποιημένη Ευρώπη σημαίνει μια κοινή κουλτούρα πρόβλεψης, προνοητικότητας και δράσης για να είμαστε μακροπρόθεσμα πιο ανθεκτικοί. Και θα ήθελα να περάσω τώρα σε συγκεκριμένα μέτρα για το πώ μπορούμε να σφυριλατήσουμε αυτή την ιδιαίτερη, την ξεχωριστή εταιρική σχέση. Φυσικά προβλέπω στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων στη φάση ήδη τη διαμόρφωση του ε, προγράμματο. Και μάλιστα θα στηρίξω την εκλεγμένη πρόεδρο για την ανάπτυξη του πρόεδρου εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι προτεραιότητά μα, γιατί το πρώτο μα πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει ήδη να συμφωνηθεί πριν το δε, ήδη από το Δεκέμβριο. Από την πρώτη στιγμή θα συνεργαστώ με του συναδέλφου Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επαφέ μαζί σα με τι πολιτικέ ομάδε και με τη διάσκεψη πρόεδρων ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με, βάση, με αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε μια κοινή διακήρυξη για τις νομοθετικές προτεραιότητες. Επίσης θα προτείνω το πρώτο πολιετές πρόγραμμα όπως προβλέπεται στην Διοργανική Συμφωνία του 2016 για καλύτερη νομοθεσία. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι μια άσκηση συνδημιουργίας με συλλογική ε, ευθύνη και λογοδοσία. Επίσης, ε, Δεύτερο, δικαίωμα πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη μια νέα θεσμική εποχή. Όπω ανήγγειλε και η εκλεγμένη πρόεδρο, όταν το Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών του απαιτεί μία νομοθετική πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανταποκριθεί υποβάλλοντα μία νομοθετική πρόταση με πλήρη σεβασμό τη αναλογικότητα, επικουρικότητα και των αρχών της καλής νομοθεσίας. Για να γίνει κάτι τέτοιο γρήγορα, θα προτείνω συμμετοχή και του Κοινοβουλίου στις ε, πρόορες φάσεις της διαδικασίας με βάση τα ψηφίσματα και συνεργασία για την διαμόρφωση αυτών των φάσεων. Επίσης, θέλω ένα μηχανισμό έγκυρης προειδοποίησης για να εξασφαλίσω συνεχή διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη στιγμή που εγκριθεί ένα, νομοθετικό, ένα ε, κοινοβουλευτικό ψήφισμα, θα εξασφαλίσω συζήτηση επί του θέματος στο συλλογικό όργανο της Επιτροπής. Και φυσικά θα πρέπει να διευκολύνουμε την κατανόηση επί της ουσίας και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων και την αίσθηση της συνεργασίας μεταξύ μας προς ένα κοινό στόχο. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, χτυπά ο παλμός της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Γι' αυτό θα συνεργαστώ με τον αρμόδιο αντιπρόεδρο για να μεριμνήσουμε ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει σημαντικό ρόλο στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και επίσης θα, θα ενθαρρύνω να αναζωογονήσουμε τις συζητήσεις για εκρεμή ε, θεσμικά ζητήματα και ιδιαίτερα το δικαίωμα εξέτασης. Επίσης, ε, θα ε, κάνουμε μία αναθεώρηση και του σχετικού κανονισμού και γι' αυτό περιμένω και με ανυπομονησία την έναρξη του τριλόγου, των τριμερών συζητήσεων. Επίσης, ό,τι αφορά τι οργανικές διαπραγματεύσεις, συνεργαστώ με τους αρμόδιους επιτρόπους ώστε να ενημερώνεται κατάλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίω πριν σημαντικές διεθνή διεθνείς εκδηλώσεις και σε βασικές ε, φάσεις διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές, είναι σημαντικές αυτές οι καταγγελίες των ε, πολιτών και θα συνεργαστώ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με την Επιτροπή Μεταφορών και φυσικά θα είμαι παρόν στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Μεταφορών. Βέβαια, ε, θα έχουμε αυτές τις αναφορές και ελπίζω να δούμε πώς θα δράσουμε ώστε να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες των πολιτών όπως, αναφέρονται σε αναφορές, όπως περιλαμβάνονται σε αναφορές. Επίσης θέλω αποτελεσματική και διαφανή εφαρμογή της ε, νομοθεσίας. Θέλω να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε διαχρονική νομοθεσία που θα αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, δεν θα δημιουργεί πλέον επιβάρηση και θα προσφέρει αποτελέσματα με ελάχιστο κόστος. Και γι' αυτό ε, θα ήθελα να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας για την ε, καλύτερη βελτίωση. Και θα ήθελα το πρόγραμμα REFIT, βελτίωση και καταλληλότητας αποδοτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου, να ανταποκρίνεται στι ε, μελλοντικέ ανάγκε στην, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τι ψηφιακέ ανάγκε. Επίση, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναμίξουμε καλύτερα του ε, δέκτε, του χρήστε τη νομοθεσία και να εφαρμόσουμε ενεργό επικουρικότητα, ώστε να μην επικρατεί εντύπωση ότι όλα αποφασίζονται στι Βρυξέλλε. Επίσης θέλουμε τοπικέ και περιφερειακές αρχές να μας ενημερώνουν για το πώς βιώνουν την γραφειοκρατική επιβάρυνση της κοινοτική νομοθεσίας και να δούμε τρόπους για να την μειώσουμε. Και περιμένω ε, ε, feedback και από εσά και σχόλια από εσά, γιατί εσεί είστε ο άμεσο σύνδεσμο μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Και σίγουρα θα εμπλέξω εδώ αποτελεσματικά και την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Επίσης θέλω καλύτερη ε, συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ώστε κατά την εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας να μην προσθέτουν περί το διοικητικό άχθος, το γνωστό κανονιστικό υπερθεματισμό, το gold plating. Επίσης θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να ενημερώνονται όταν τα κράτη-μέλη θεσπίζουν επιπλέον και περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Θα φροντίσω ώστε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνονται κατάλληλα επίσης για αυτό το θέμα. Τα πρώτα δύο χρόνια της θητείας μου σκοπεύω να επισκεφτώ όλα τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια που εκτιμώ τον ρόλο τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενεργό επικουρικότητα και αναλογικότητα και θα ζητήσω μαζί στον πολίτη προγραμματισμό και θα εφαρμόσω την αρχή ένα μπαίνει, ένα βγαίνει, one in, one out, που ανήκει η εκλεγμένη πρόεδρος. Δηλαδή για κάθε νέα νομοθετική πρόταση με νέα επιβάρυνση για τους χρήστες θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται ισοδύναμη ελάφρυνση αντίστοιχη ε, επιβάρυνση αλλού. Και αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. και θα ήθελα η νέα αρχή να εφαρμοστεί σε όλου του τομεί. Βέβαια και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, Λέω ένα κατηγορηματικό όχι σε μια μηχανική προσέγγιση και στην υπονόμευση ή διακύβευση των υψηλών μας προδιαγραφών, ιδιαίτερα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταθμίζουμε και τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επιτελέσει εξαιρετικό έργο με, το, με τη μελέτη για το κόστο τη μη Ευρώπη. Ποσοτικοποίησε το οικονομικό κέρδο σε 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ για μία δεκαετία. Αν, για παράδειγμα, εφαρμόσουμε πλήρω την ενιαία αγορά και κυρίω στι επιχειρήσει, τον ψηφιακό τομέα, την ενέργεια και αν ε, διορθώσουμε το θέμα της φοροαποφυγής από τις επιχειρήσεις. Και μέσω της σύνοψης ε, και της ενωτικής ενημέρωσης για τους πολίτες θα ήθελα να γίνεται καλύτερη επικοινωνία και για τα τεκμηριωμένα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτες, επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικώ. Επίσης, ε, θα πρέπει να επιτύχουμε σε διοργανικό επίπεδο, κάτι που είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχή πολιτική. Θα πρέπει να τα συνδέσουμε όλα αυτά και αυτό θα φέρει ρηξικέλευτε αλλαγέ που δεν είναι καθόλου αφηρημένε. Για παράδειγμα, έχουμε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για του Σορευτέ ακόμη και την τελευταία στιγμή καταφέραμε να προλάβουμε τις τεκτονικές αλλαγές προς την ηλεκτρονική κινητικότητα και μάλιστα με ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας ξεκινήσαμε μια στρατηγική δράση για να δημιουργήσουμε μια αξιακή αλυσίδα και να ξεκινήσουμε την παραγωγή φιλοπεριβαλλοντικών συσσωρευτών εδώ στην Ευρώπη. Και έτσι καλύπτουμε το έδαφος με τους Ασιάτες ανταγωνιστές μας για ένα βιώσιμο μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανία μας στην Ευρώπη που φαίνεται πια διασφαλισμένο και με τιμά ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εκλεγμένη πρόεδρος ε, μου ανέθεσε τα θέματα αυτά και την, τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης και σε συνεργασία με άλλους στρατηγικού τομείς πραγματικά θα κάνουμε τη διαφορά αρκεί να συνεργαστούμε και γι' αυτό αν μου δώσετε την έγκρισή σας θα προτείνω να προσπαθήσουμε να έχουμε μια παγκόσμια κλάση σε προνοητική διακυβέρνηση και με ιδιαίτερε ικανότητε διορατικότητα και πρόβλεψη εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Επίση, θα κινητοποιήσω του πόρου του Κοινού Κέντρου Ερευνών που είναι σημαντικό ε, φορέα και παράγοντα. Επίση, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο στρατηγική πρόβλεψη που θα αξιοποιήσει στο έπακρο το καλύτερο δυναμικό των κρατικών ε, και θεσμικών οργάνων. Φυσικά, ο καθένα ε, έχει τις απόψεις του, αλλά θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των δράσεών του. Και απέναντι σε αυτή την παλήρη των πληροφοριών θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ποιότητά τους και να ενισχύσουμε τη διαφάνειά τους. Θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι τεκμηριωμένες. Και επίσης θα προσπαθήσω να συστήσουμε ένα κοινό μητρό τεκμηρίων ανοιχτό στο κοινό που θα περιλαμβάνουμε την τεκμηρίωση που χρησιμοποιούμε στις νομοθετικές μας προτάσεις. Όπως ξέρετε, η κυρία Ούρσουλα Φοντερ μου είπε ότι θα πρέπει να ετοιμάζω ετησίως μια έκθεση προβλέψεων για τις αναδυόμενες τάσεις και θα αναφέρεται και στις προγραμματικές μας ε, συζητήσεις θα πρωτοστατήσω σε στρατηγικές συζητήσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θέλω να συμφωνήσουμε για κάποιες ε, ε, μέγα τάσεις που θα φέρουν επαναστατικές αλλαγές και θα μας επηρεάσουν στη στρατηγική μας προσέγγιση και θα επηρεάσουν επίσης άμεσα και τον πολιτή μας προγραμματισμό. Με όλα αυτά κατά νου θα συνεργαστώ στενά με τον Αντιπρόεδρο, τον, Αρμόδιο, στα πλαίσια της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είχα την τιμή να συνεργαστώ με τις δικές σας ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές στη διάρκεια της περασμένης θητείας, κυρίως και πάνω απ' όλα με την Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, καθώς και με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, στη συνέχεια με την Επιτροπή Έρευνα, ε, Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, ώστε να δημιουργήσουμε την Ένωση Ενέργειας. Στην πρώτη μου θητεία ολοκληρώσαμε τη Συμφωνία Πλαίσιο ανάμεσα στα θεσμικά μας όργανα Εργαστήκαμε χέρι με χέρι για να επιτύχουμε τον εξυγχρονισμό του καθεστώτων των υπαλλήλων και άλλων ε, συνεργατών. Ε, συνεργαστήκαμε για να θεσπίσουμε κοινούς στόχους. Στόχος μου είναι να, να εργαστώ ακούραστα ώστε να επιτύχω τους στόχους μας, ε, καθώς εμπνέομαι από τους δημοκρατικούς, ε, δημοκρατικές αξίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς. Ξεκινάμε με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Πρώτη ερώτηση θα τεθεί από τον κύριο Βοσ, που είναι συντονιστής του ΕΛ και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Σεφτσοβιτς. Έχω την τιμή να κάνω την πρώτη ερώτηση για να ελαφρύνει ο γραφειοκρατικός φόρτος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ε, θα κάνετε καμιά προσπάθεια ε, για να το ελαφρύνετε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάτε για την αρχή one in, one out. Πώς θα γίνει αυτό και πώς ε, θα εφαρμοστεί συγκεκριμένη η αρχή έτσι ώστε να αποφεύγεται ο άχρηστος γραφειοκρατικός φόρτος και πότε να αναμένουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ ένα τέτοιο μέσο. Απάντηση. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή κύριε Φως. Πρώτον, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και πάρα πολύ σοβαροί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε συναντήσει ε, όλοι δυσαρεστημένους πολίτες και επιχειρηματίες που μας λέγουν ότι είναι ακρεφνείς υποστηρικτές της Ευρώπης, αλλά διστάζουν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση γιατί τους τρομάζει αυτό το γραφειοκρατικό άχθος και χαίρομαι που η εκλεγμένη πρόεδρος θέλει να δώσει εκεί έμφαση τη μείωση ε, των άχρηστων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ε, πάντως θα πρέπει ε, αυτή η αρχή να μην εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση μηχανικά και αυτόματα και ούτε να μειώσουμε τις ε, ε υψηλές προδιαγραφές που έχουμε για το περιβάλλον ή για τα κοινωνικά ζητήματα. Πώς θα το κάνω αυτό θα αλλάξω το πρόγραμμα REFIT και θα το μετονομάσω σε Fit for the Future, ε, έτοιμη για το μέλλον. Ε, παραδοσιακά γίνεται μια αξιολόγηση για το πώς αποδίδει η νομοθεσία. Αυτό είναι το REFIT, αλλά και αυτό χρειάζεται αναβάθμιση. Είναι αρκετά ψηφιακή, ε, συνάδει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή government. Πλησιάζει πρώτα τους μικρούς. Υπάρχει φόρτος αυτός ο νομοθετικός είναι, έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή με τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία. Ή έχει να κάνει με το τελευταίο παράρτημα, το τελευταίο πίνακα σε μια νομοθετική πράξη που πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η προσέγγιση μας για να βεβαιωθούμε ότι ακόμα και όταν εγκρίνουμε νέα νομοθεσία που χρειάζεται πάντα να έχουμε υπόψη μας πώς μπορούμε να το κάνουμε και πώς να εστιάσουμε ε, για να υπάρχει αυτή η πειθαρχία σε όλα τα θεσμικά όργανα που θα έχουν πάντα υπόψη την ανάγκη ε, μείωσης ε, του γραφειοκρατικού άχθους που προκαλούν σε κάποιους άλλους. Ευχαριστώ. Είστε ικανοποιημένο, κύριε Φως. Πολύ ωραία. Δεύτερη ερώτηση είναι από τον κύριο Πέντρο Σίλβα Περέιρα, σοσιαλιστές και δημοκράτες στην ΑΦΚΟ. Συντονιστής. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε και υποψήφιε Επίτροπε. Καλώς ορίσατε στο σώμα αυτό. Το γνωρίζετε ήδη καλά γιατί ασκείτε καθήκοντα Επιτρόπου από το 2009 και έχετε την ευθύνη για τις διαθεσμικέ σχέσεις και άρα λοιπόν αυτό μας δίνει ε, λαβή για αισιοδοξία για τις σχέσεις μεταξύ μας. Για τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης χρειαζόμαστε ένα Ευρωκοινοβούλιο με ενισχυμένο ρόλο αυτό που θέλω να σας ε, ρωτήσω είναι πώς η συμμετοχή ε, του Ευρωκοινοβουλίου θα γίνει για τη, στη μελλοντική συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλουμε να έχουμε μια δραστήρια συμμετοχή ε, και ηγετική θέση ή απλώς σκοπεύετε να μας καλέσετε ως τιμόμενο πρόσωπο. Έπειτα, το Ευρωκοινοβούλιο τηρεί τους, ε, τις διαθεσμικές συμφωνίες που ήδη ισχύουν, ειδικά αυτό που ισχύει για την ε, οικονομική διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, πώς μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά. Σας ευχαριστώ και εκτιμώ τις ερωτήσεις από του συναδέλφου Περέιρα. Καταρχάς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα δύο κοινοτικά ε, θεσμικά όργανα ε, όχι μόνο θα ε, βασιστούν σε μια ιδιαίτερη σχέση, αλλά θα συνεργαστούν πιο στρατηγικά για το κοινό μας μέλλον. Πιστεύω πως το Ευρωκοινοβούλιο θα ήταν το κατάλληλος χώρος για να συζητηθεί το μέλλον της Ευρώπης ακόμα και μετά από τη δική μας θητεία. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι αποφασίσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια πραγματικά θα χαράξει την, θέση της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια. Και αν ήθελα να είμαι πιο ε, δραματικός, πιστεύω πως τώρα αποφασίζεται το πρόσωπο της Ευρώπης για ολόκληρο τον αιώνα αυτό. Τα όσα αποφασίζουμε λοιπόν θα παίξουν χαρακτηριστικό ρόλο, αποφασιστικό ρόλο για το θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει βασικό ρόλο. Ε, τώρα, ερχόμενοι πιο κοντά στις καθημερινές μας σχέσεις όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Εδώ σαφώς θα πρέπει να συνεργαστούμε και η υποψήφια πρόεδρος ήταν σαφής ότι είναι έτοιμη στο να συνεργαστεί στενά με το Ευρωκοινοβούλιο και να δεχτεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο και, τα μέλη, και, μάλλον, και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ηγηθεί αυτή τη διάσκεψη. Πιστεύω πως επίσης αυτό που το τονισέ ήταν το γεγονός ότι αυτή η διάσκεψη θα πρέπει να βγει και κάπως εκτός των ε, τυχών των Βρυξελών. Να πάμε δηλαδή στους πολίτες κοντά, στις πρωτεύουσε, να συνομιλήσουμε μαζί τους, να καταλάβουν ότι πραγματικά γνωρίζουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και αν ε, μπορέσουμε με επερώτηση και για τις διαθεσμικές σχέσεις θα επανέλθω ε, σε επόμενη ε, και θα συμπληρώσω. Εσείς είστε ικανοποιημένος κύριε Περέιρα. Ναι, Υπάρχει χρόνος από ό,τι κατάλαβα. Ε, θα ήθελα πραγματικά να δώσουμε την ευκαιρία στον ε, κύριο υποψήφιο επίτροπο για να αναφερθεί στο θέμα της εφαρμογής των διαθεσμικών συμφωνιών που μάλιστα τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί εκείνος διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία πλαίσιο του 2010 και που αποτελούν αυτές οι συμφωνίες το θεμέλιο της σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θυμάμαι τις πολύ δυναμικές διαπραγματεύσεις που κάναμε το 2009 και είμαι ευτυχής που η Συμφωνία Πλαίσιο άντεξε στη δοκιμασία του χρόνου, αλλά θυμάμαι ότι και τότε προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κομμάτι της, ε, της ε, Συμφωνίας Πλαίσιο. Δηλαδή, στόχος ήταν να λισαβονοποιήσουμε τις σχέσεις μας και πιστεύω πως αν κατάλαβα αν, και αν έχω την έγκρισή σα, θα έχω αυτή την προσέγγιση προ το Συμβούλιο πάλι. Θα του πω έχουμε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, Α την εξετάσουμε, Α δούμε τι πρέπει να εξυγχρονιστεί και να μπορέσουμε να κάνουμε το Συμβούλιο να συνεργαστεί πιο στενά μαζί μα και επί τη βάση αυτή τη συμφωνία. Το καταφέραμε αυτό στη συμφωνία για την καλύτερη ε, νομοθεσία. Πιστεύω πω μπορούμε να το επιτύχουμε και με αυτή την συμφωνία πλαίσιο. Ο τρίτο συντονιστής, η συντονίστρια της Τουρινιού στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η Κάρεν Μελχιόρ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε που ήρθατε εδώ. Μου άρεσε η αρχική σας δήλωση ε, που θέλετε τεκμηριωμένη και διαχρονική νομοθεσία που θα αντέχει δηλαδή στη δοκιμασία του χρόνου και μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα συμβάλλει σε αυτό. Η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω για την καλύτερη νομοθεσία επικρίθηκε γιατί δεν έλαβε δεόντω υπόψη το κίνδυνο επιπτώσεων, ε, τον αντίκτυπο ε, των μέτρων ή την επιλεκτική δημοσίευση ή μη δημοσίευση κάποιων τέτοιων μελετών και μέτρων. Για παράδειγμα, για κάποιες τεκμηριώσει που έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ε, είχαν γίνει κάποιε κοινέ αναλύσει με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια πορίσματα επιστημόνων τη επιστημονική κοινότητα. Πώ θα μεριμνήσετε ώστε όλα τα επιστημονικά πορίσματα, όλη η επιστημονική τεκμηρίωση και η μελέτη επιπτώσεων θα περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρό που αναφέρατε και θα είναι προσιτέ στο κοινό υποψήφιο επίτροπο Ευχαριστώ κυρία μου για την ερώτηση και θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερο την εμπειρία που είχαμε για τον τρόπο εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη δυνατότητα εξυγχρονισμού τη της Και μάλιστα την δανεική ε, ε, τη Δενική Ένωση Επιχειρηματιών και τα σχόλιά τους. Σε ό,τι, αφορά, την ανάγκη διαχρονικότητας της μελλοντική μας νομοθεσίας, νομίζω ότι το βασικό στοιχείο της θα είναι ε, να ανταποκρίνεται στις ανάγκε των καιρών και από ψηφιακή άποψη, δηλαδή να αποφύγουμε κάποιες ε, στο φαξ, γιατί όταν ε, με ρώτησαν κάποιοι τι φάξ, τι θα πει φάξ, τι μηχάνημα είναι αυτό. Και παρόλα αυτά υπάρχει ακόμη σε κάποιες νομοθετικές ε, προτάσεις και διατάξεις. Θα πρέπει λοιπόν από ψηφιακή του άποψη να είναι εξυγχρονισμένα τα νέα μέτρα και αν δεν είναι να τα εξυγχρονίσουμε. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο ε, των μέτρων και μια τεκμηριωμένη νομοθεσία, θα πρέπει και εδώ να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τις μελέτες επιπτώσεων και την τεκμηρίωση. Πραγματικά ε, εκπλήσωμε από τον όγκο των πληροφοριών που έχουμε στα θεσμικά μας όργανα και στο Κέντρο Κοινών Ερευνών. Και, και η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και οι αντίστοιχε ε, μονάδες και τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεργάζονται στην εκπόνηση τέτοιων μελετών. Είχατε τη δική σας πολύ αξιόλογη μελέτη για το κόστος της μη Ευρώπης. Θα ήταν κρίμα να αποκρύπτουμε αυτές τις πληροφορίες ή να τις κρατούμε ε, μόνο για τον εαυτό μας. Η ιδέα μου λοιπόν είναι να συστήσω ένα διοργανικό μητρό ε, στην οποία θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση και όλη η εργασία που έχει γίνει και οι μελέτε των επιστημόνων και τα επιστημονικά πορίσματα θα είναι διοργανικού χαρακτήρα το μητρό αυτό, υπό το δικό σα λοιπόν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και εκεί θα περιλαμβάνονται όλε αυτέ οι τεκμηριωμένε επιστημονικέ μελέτε που θα αποτελέσουν τη βάση για την μελλοντική εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων. Είστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ για την απάντησή σας κύριε Επίτροπε, ε, υποψήφια Επίτροπε. Προσβλέπω σε ένα πιο ανοιχτό και διαφανές μητρό τεκμηρίωσης και ελπίζω η μελλοντική μας ε, νομοθεσία να είναι πραγματικά διαχρονική και από την άποψη της ψηφιοποίησης και των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Έχουμε και το θέμα τώρα της ανάμειξης της εμπλοκής των Ευρωπαίων πολιτών που θα είναι θεμέλιο της καλύτερης νομοθεσίας. Και η επιρροή του στη διαμόρφωση νομοθεσίας θα έχει κέρια θέση για την ε, δημοκρατία μας. Σε μια πρόσφατη υπόθεση είχαμε την ε, δεδηλωμένη ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών για κάποιες πτυχές της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι, οι Ευρωπαίοι πολίτες έκριναν ότι αγνοήθηκαν ε, και παραμερίστηκαν οι, οι απόψεις τους και μάλιστα ε, μερικέ φορέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιφρονητικά αναφέρθηκε στι απόψει αυτέ, χαρακτηρίζοντα τι bots και ότι δεν ήταν ουσιαστικέ ε, προτάσει. Πώ θα φροντίσετε ότι στο μέλλον να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανησυχίε και οι προτάσει των Ευρωπαίων πολιτών. Σα ευχαριστώ για τι πολύ εύστοχε ερωτήσει σα. Πιστεύω ότι όλοι μα θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια πιο ευρυθή ανάλυση του τι μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία και με την ε, Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με τις ε, τρεις επιτροπές, την ΑΦΚΟ, τη Γιούρη και την Επιτροπή Αναφορών. Επίσης, μερικές φορές οι πολίτες ε, αποθαρρύνονται για συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις και ε, μπορεί να είναι καλή διοργάνωση, αλλά μερικά είδη διαβουλεύσεων ίσω ε, μπερδεύουν του Ευρωπαίου πολίτε. Οπότε, αν θέλουμε περισσότερη και καλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στι δημόσιε διαβουλεύσει, θα πρέπει να τι ε, διαφημίζουμε καλύτερα. Δηλαδή να συνεργαστούμε με επαγγελματικέ ενώσεις, συλλόγους, με οργανώσεις νεολαίας, με τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διάφορες πρωτεύουσες Να μην γίνονται όλα από τις Βρυξέλλες να έχουμε πιο στοχοθετημένε συζητήσεις με τους πολίτες Και αυτό που περιμένουν κυρίως οι πολίτες είναι μια απάντηση από εμά, μια ανταπόκριση. Να καταλαβαίνω ότι κάποιο εξετάζει τις απόψεις τους τις αξιολογεί, τις σταθμίζει και εκτιμά τη δική του συμβολή. Επόμενη ερώτηση από τους Πρασίνους. Ο κύριο Ντάνιελ Φρόιντ έχει το λόγο συντονιστή στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Σεύτσοβιτς, ευχαριστώ που ήρθατε να απαντήσετε σήμερα στι ερωτήσεις μας. μέτρησα ε, τι προτάσεις ε, στι επιστολέ ανάθεση χαρτοφυλακίων ε, των συναδέλφων σα 97 προτάσει για νέα νομοθεσία και εσεί καλείστε να μειώσετε τη γραφειοκρατία με αυτό το σύστημα one in, one out. Ε, τι θα διαγράψετε από αυτές τις 97 προτάσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Θα έρθει το μεγάλο πακέτο για το κλίμα που έχει εξαγγελθεί ε, μέσα στις πρώτες 100 μέρες. Μήπως να ανησυχούμε ότι θα επανέλθει η περιαγωγή. Το θέμα δεν είναι ποσοτικό, πόσους νόμους θα αλλάξουμε. Αυτό που ενοχλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι ότι αν θέλει κανείς να πάρει μια μικρή υποτροφία για το Εράσμους, έχει ένα βουνό ε, διατυπώσεις να κάνει και ε, έντυπα να συμπληρώσει. Μήπως να μειωθούν τα έντυπα, αντί να μειώνονται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές ή κοινωνικές, ε, τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα. Ο Αντιπρόεδρος Σεύσοβιτς, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για την τόσο έντονη δήλωση και στεναρή, την οποία συμμερίζομαι. Θα ήθελα να διαβεβαίωσω και τους βουλευτές και τους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν ε, για τις υψηλές προδιαγραφές και πρότυπα έχουμε, είτε αυτά είναι κοινωνικά είτε περιβαλλοντικά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα βελτιώνουμε συνέχεια. Τι θέλει να κάνει η εκλεγμένη πρόεδρος στην προσέγγιση αυτή, one in, one out μια νέα πειθαρχία για το πώς θα κοιτάξουμε το γραφειοκρατικό άχθος αυτό. Όταν φέρνουμε ένα νομοθέτημα ε, θα πρέπει να δούμε ε, πόσο θα επιβαρύνει περισσότερο τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους μικρομεσαίους και πού μπορούμε για κάθε νέα νομοθεσία να φέρουμε μια παλιά. Ε, αν είναι απαρχιωμένη, αν χρησιμοποιεί το φαξ ή τα χαρτιά και μπορούμε να τη βελτιώσουμε, να την κάνουμε ταχύτερη, πιο ενημερωμένη και πιο σύγχρονη και πιο φιλική προς τον πολίτη από ό,τι είναι μέχρι σήμερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά μας των πρώτων 100 ημερών για το νέο πράσινο deal, για τον κατώτατο μισθό, για τη διαφάνεια στις αμοιβέ. Θέλουμε να έχουμε ήδη αποτελέσματα. Και επίσης θέλουμε και νέους κανόνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ε, θα έχουμε και μία προσέγγιση Ε, απέναντι στο γραφειοκρατικό φόρτο πάρα πολύ ε, λογική, με πολύ μεγάλη ευαισθησία και σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε εκπτώσεις ε, στις απαιτήσει μας. Ε, όπως γνωρίζετε θα πρέπει να ε, αποφασίσουμε και όλα, για όλα τα νομοθετήματα που εκκρεμούν, που είναι ακόμα ε, επιτάπητος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πάνω από 100. Θα πρέπει να μελετήσουμε συλλογικά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτούς τους φακέλους, αλλά θα ενημερωθείτε δεόντως και γέρος. Είστε ικανοποιημένος από την απάντηση. Ε, θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, μιλάτε πάντα για στοιχεία και για πολιτική που να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα πρέπει να εδράζεται σε επιστημονικά θεμέλια. Έχουμε 26.000 όμως επιστήμονες στην Ευρώπη που λένε ότι η σημερινή πολιτική για το κλίμα δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα και έκτακτη ανάγκη που έχουμε για το κλίμα. 1033 είναι τα νομοθετήματα από το 1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επόμενη πενταετία θα τα τσεκάρετε αυτά αν συνάδουν με τη Συμφωνία του Παρισιού και όλα τα νέα νομοθετήματα που επίκυνται. Ε, για να το μεταφράσω αυτό στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μελέτες αντικτύπου, αυτό το impact assessment, μήπως πρέπει να αλλάξει εκβάθρον ο τρόπος που γίνονται και να μην φτάσουμε στον 1,5 βαθμό Κελσίου αύξηση πριν τελειώσει η θητεία σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή επίσης. Γίνεται αυτό το καιρό μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία αντανακλάται πάρα πολύ και στη δική μας περισυλλογή ε, για το πώς θα αλλάξουμε αυτές τις μελέτες αντικτύπου ε, τις περιβαλλοντικές. Ε, θα πρέπει να βάλουμε περισσότερο υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία. Αρκούν αυτά που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Μετράμε αρκετά τον κοινωνικό αντίκτυπο. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία ποιον εξυπηρετεί. Αντέχει στο χρόνο και τις ε, αλλαγές, τις ε, μόνιμες. Πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αυτές τις μελέτες αντικτύπου και αυτό θα το συνδυάσουμε με τις προβλέψεις για να κοιτάξουμε πώς ε, ε, φανταζόμαστε την Ευρώπη μετά από 10-20 χρόνια και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν δημοσιεύουμε ε, σε αυτό το κοινό μητρό όλα τα στοιχεία και όλα τις νομοθεσίες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ζηρόμ Ριβιέρα, εξ ονόματος της ομάδας ΙΔΕ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεφτσοβίτς, ε, καλημέρα σας ε, και σας θέτω την ερώτησή μου εξ ονόματος της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία και το διευκρινίζω γιατί έχουμε γίνει αντικείμενο πολύ άσχημης μεταχείρισης. Ο νόμος don't συστηματικά μας έχει απαγορευθεί και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στα διάφορα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι μέτρα λοιπόν θα λάβετε θα, ε, στην Επιτροπή ώστε να ακούσετε την φωνή των ερετών ε, που οι βουλευτές ε, στην χώρα μας ήρθαν επικεφαλής στις λίστες, στα ψηφοδέλτια. Επίσης, έτσι εμφισβητούνται τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Ας πούμε, στη Γαλλία συζητήθηκε διάφορα θέματα. Ποια μέτρα προβλέπετε για να μπορέσει η κοινωνία μας να προχωρήσει σε δρόμους που εξασφαλίζουν και κοιώνται τα συμφέροντα τα ατομικά αλλά και τα συλλογικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Η Κομισιόν ως θεματοφύλακας των συνθήκων θα πρέπει να είναι στενός συνεργάτης του Ευρωκοινοβουλίου. και οι μεταξύ μας ανταλλαγέ απόψεων θα περιέχουν καλές συμβουλές που θα εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Θα αναζητήσουμε ε, δρόμους για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με όλες τις ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Πιστεύω πως χρειάζεται να αναπτύξουμε και νέες μεθόδους. Μιλούσα για τη δημόσια διαβούλευση, για τα διάφορα επίπεδα της ανταπόκρισης που έχουμε όταν ε, ας πούμε ε, συζητάμε. Έχουμε 4,6 εκατομμύρια άνθρωπους που μας γράφουν και μας λένε ότι θέλουν να ε, συμμετέχουν στο σύστημα. Να σε άλλες περιπτώσεις έχουμε λιγότερο ενθουσιασμό και απαντήσεις και αυτό συμβαίνει γιατί ο κόσμος δεν ενημερώνεται πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το τι προετοιμάζουμε και πώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι δημόσιες διαβουλεύσεις να διαδίδονται περισσότερο στις χώρες μας μέσω από ενώσεις αλλά και με τη δική μας προσπάθεια ώστε να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στο μέλλον. Και όσον αφορά τις μελλοντικέ τεχνολογίες νομίζω πως το... η πρώτη δοκιμή θα γίνει πολύ πολύ σύντομα και θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η GDPR θα είναι στο ύψος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πώς θα μεταφραστεί με τις νέες ε, ψηφιακές τεχνολογίες. Πώς λοιπόν ε, θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αντικατασταθούμε από τους ε, μηχανές. Ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε περώτηση. όσον αφορά το σεβασμό του Κοινοβουλίου, ποια είναι η θέση σας απέναντι σε μια διαδικασία που θα άξιζε κόκκινη κάρτα, που θα επέτρεπε δηλαδή να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Εάν δηλαδή μια πλειοψηφία βουλευτών απορρίψει μια πρόταση της Κομισιόν του Κοινοβουλίου, να μπορούμε να έχουμε αυτό το δικαίωμα βέτο για να προχωρήσουμε περισσότερο και να γίνει έτσι σεβαστή και η ε, εθνική κυριαρχία και τα εθνικά κοινοβούλια. Και πάλι εδώ θα είμαι πολύ ε, πρακτικός. Πολύ συχνά συνομιλώ με τα Εθνικά Κοινοβούλια και γνωρίζω πόσο πολύ σημαντικό είναι, πόσο σημαντικές είναι οι κίτρινες κάρτες, οι πράσινη κάρτα και οι κόκκινες κάρτες είναι πολύ παρούσες στη συζήτησή μας. Επίσης, αυτό που, εξηγώ, που εξηγούσα στους συναδέλφους και ε, είμαι έτοιμος να το επεξεργαστώ περισσότερο από πολιτική άποψη είναι ότι όταν ας πούμε στην Κομισιόν δούμε ότι η πρόταση που είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε θα αντιμετωπίσει αντίθεση, αμφισβήτηση από πάνω από το 50% των Εθνικών Κοινοβουλίων, δεν θα τη θέσουμε επιτάπητος. Είμαστε ρεαλιστές. Εφόσον έχουμε την αντίρρηση άνω του 50% των Εθνικών Κοινοβουλίων, δεν θα εγκριθεί. Επίσης υπάρχουν καλά παραδείγματα για την πράσινη κάρτα. Όταν ας πούμε πήραμε τις επιστολές από, παίρνουμε τις επιστολές από τα εθνικά κοινοβούλια ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα με τα απόβλητα τροφίμων. Ε, τα, κάνα, τα πήγαμε καλύτερα, κάναμε τις προτάσεις για την κυκλική οικονομία και τα εθνικά κοινοβούλια είναι ευχαριστημένα με το πόσο γρήγορα αντιδράσαμε. Χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία λοιπόν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεργαζόμαστε στενότερα με τα εθνικά κοινοβούλια. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Άγγελ Τζαμπάτσκι από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την Ομάδα Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επιτροπέ, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για το μέχρι τώρα σας έργο και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια. Θα ήθελα να συνεχίσω τον ερμό του προλαλήσαντα. Θα αρμόδιος και για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και επίσης αρμόδιος για την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της επικορικότητας και τους δεσμούς ε, με τους βουλευτές που εξυπηρετούν ε, τους που υπηρετούν και προσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων, ιδιαίτερα στα θέματα επικορικότητα και αναλογικότητα. Τι συγκεκριμένα θα προτείνετε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κίτρινη και πορτοκαλί κάρτα. Και επίσης, τι θα κάνετε με την αρχή one in, one out. Για μια νέα, κάθε νέα επιβάρηση, ισοδύναμη επιβάρηση θα φερείτε διοικητικά. Η νέα αυτή αρχή, one in, one out, πώς θα εφαρμοστεί ακριβώς Επίσης, θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρότερο ρόλο και μεγαλύτερη ανάμειξη των ενδιαφερομένων και ενεχομένων, δηλαδή των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Σεύτσοβιτς, έχετε το ρόλο. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκη για την ερώτησή σας. Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα εξέτασα με μεγάλη προσοχή και Μία ιδιαίτερα ιδέα χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και επεξεργασίας η έννοια της ενεργούς ε, επικουρικότητας. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε στην ευρωπαϊκή συζήτηση να συμπεριλάβουμε και τα εθνικά κοινοβούλια τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ και τι περιφερειακές βουλές αν υπάρχουν και μάλιστα σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, ώστε να ε, νιώθουν ότι είναι τμήματα της ευρωπαϊκής προσπάθειας και να μπορέσουν να διατυπώσουν ε, τι ανησυχίε του για τη διοικητική διατύπωση ή προβλήματα εφαρμογής σε συγκεκριμένη περιφέρεια, σε συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η προβληματα εφαρμογη σε συγκεκριμενη περιφερεια σε επικουρικότητα θα εξασφαλίσει τη διαχρονικότητα της νομοθεσίας μας και την μεγαλύτερη αποδοχή της και την καταλληλότερη και πιο σωστή εφαρμογή της. Γιατί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε με τη γραφειοκρατία είναι ακριβώς αυτός ο κανονιστικός υπερθεματισμός, αυτό το gold plating. Όταν δηλαδή κάποια περιφερειακά ή εθνικά κοινοβούλια προσθέτουν κατά τη μεταφορά της ε, οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο νέα στοιχεία, νέες επιβαρύνσεις που καθιστούν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου πολύ πιο περίπλοκη. Εκτιμώ ιδιαίτερος ε, το έργο που έχει επιτελέσει το θέμα αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών και την ανάπτυξη κάποιων περιφερειακών κόμβων, ένα δίκτυο των περιφερειακών αρχών ώστε να ενημερωνόμαστε κατάλληλα για τα προβλήματα που υπάρχουν και να μπορέσουμε εγκαίρως να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δίκτυο θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες διαβουλεύσεις, Θεωρώ τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, η διαβούλευση με τις επαγγελματικές ενώσεις, είναι πολύ χρήσιμες διαβουλεύσεις, μαθαίνουμε πολλά από αυτές και έτσι θα διευκολύνουμε και την κατάλληλη αντίληψη για το, για το ευρωπαϊκό δίκαιο και την καλύτερη εφαρμογή και αποτελεσματικότερη μεταγραφή του στην εθνική νομοθεσία. Τώρα, ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ, συντονιστή ε, στην ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Σεφσουβίτς. Επανέρχομαι στο δικαίωμα πρωτοβουλίας και ε, στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συγκεκριμένα και σε σχέση με τη διάσκεψη που επίκειται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις νομοθετικές προτάσεις και πώς θα συμμετέχουν εκεί ε, ενεργά οι πολίτες και πώς θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη έχοντας δικαίωμα λόγου και ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη δεύτερη ερώτηση για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτς. Πολύ εύστοχα τα ερωτήματά σας, γιατί αν θέλει κανείς να, να πετύχει αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, πραγματικά θα πρέπει να τη φέρει πιο κοντά στους πολίτες μας. Yeah. Όπως είπα και προηγουμένως, πριν από λίγα λεπτά, αυτή τη συζήτηση δεν την κάνω μόνο εδώ, ε, ε, θα πρέπει να γίνει εδώ στο Στρασβούργο ή στις πρωτεύουσές μας, αλλά και στην περιφέρεια να φτάσει μέχρι τους πολίτες. Έχω αρκετή εμπειρία με ε, το διάλογο με τους πολίτες και προετοιμάζοντας τη σημερινή ακρόαση ξαναδιάβαζα κάποια στοιχεία και ξανά βλέπα από το διάλογο με τους πολίτες. Ε, ήρθαμε σε επαφή όλοι οι επίτροποι με αυτούς τους διαλόγους με 200.000 πολίτες. Ε, από δίδυ, λοιπόν, ξέρουμε πώς να φτάσουμε μέχρι τους πολίτες και τι διδάγματα αντλήσαμε από εκεί. Ότι θα πρέπει να φέρουμε στη συζήτηση τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερα περιφερειακού, τοπικού ενδιαφέροντος ή κάτι που έχει να κάνει μια συγκεκριμένη ε, βιομηχανία σε μια περιφέρεια ή κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για την νεολαία. Ε, που, τους νέους που ρωτάνε τι να σπουδάσουν για να έχουν μέλλον και μια δουλειά στην Ευρώπη και να μπορούν να είναι χρήσιμοι πολίτες, να συνεισφέρουν στην κοινωνία και να είναι προετοιμασμένοι για την όλο και πιο δυναμική αγορά εργασίας. Επίσης έμαθα ότι αν θέλεις να κάνεις μια καλή συζήτηση, καλό είναι να έχεις κάποιον που χαίρει γενικής αποδοχής στην περιφέρεια του μαζί σου στο Προεδρείο. Ε, πολλές φορές είχαν έρθει βουλευτές, ε, ευρωβουλευτές όπως εσείς ε, μαζί μου και ήταν πολύ καλή εμπειρία. Άλλες φορές ε, ε αιρετοί άρχοντες, δήμαρχοι. Είναι πολύ καλό να συνδέουμε αυτές τις συζητήσεις με το τοπικό στοιχείο παντού στην Ευρώπη ε, και να φτάζουμε όσο γίνεται σε περισσότερους πολίτες με θέματα που τους ενδιαφέρουν. Και πάντα οι συμβουλές σας και η εμπειρία σας από τις δικές σας εκλογικές περιφέρειες θα είναι πολύτιμες. Είστε ικανοποιημένο κύριε Σόλτς. Συμπροματική ερώτηση. Αυτό τι σημαίνει. Ποιος είναι η κινητήρια δύναμη αυτής της εξέλιξης. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε, δικαιολογούμαστε, νομιμοποιούμαστε να συνδιαμορφώνουμε εκεί το πρόγραμμα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω και με το Συμβούλιο. Και ε, η αρχή αυτό του one in, one out Δηλαδή για κάθε νομοθεσία που έρχεται ε, να αποσύρεται μια άλλη ε, είναι ο σωστός τρόπος ή είναι προθύστερο. Για την πρώτη περίπτωση. Ε, αν ρωτάτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα εμεί χαιρόμαστε να έχουμε το δικαίωμα πρωτοβουλία, αλλά εδώ συζητούμε για τη συμμετοχή των πολιτών στι εκλογικές σα περιφέρειες και εδώ πραγματικά θα ήταν πολύ καλό το εγχείρημα. Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος που προετοιμάζει αυτή τη διάσκεψη ε, είμαι βέβαιος ότι θα έρθει σε εντατικές επαφές μαζί σας και με χαρά να συμμετέχω κι εγώ για να ε, δώσω και τη δική μου εμπειρία Τώρα αρχίζουμε και συζητάμε τον πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό της προβλέψης, τις νέες αναδυόμενες τάσεις και όταν θα έρθει η ώρα της συγκεκριμένης ε, φαντάζομαι ότι θα βρούμε ε, ένα μοντέλο που θα ενδιαφέρει και όλους τους πολίτες και θα συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης. Και για τη δεύτερη ερώτησή σας φυσικά η αηφορία θα πρέπει να είναι ε, και η βιωσιμότητα στοιχείο κάθε μελέτης αντικτύπου και κάθε κίνησης που θα κάνουμε στην νομοθεσία. Thank you very much. Now... Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τώρα το δεύτερο γύρο ερωτήσεων, τις οποίες θέτουν τα μέλη των διαφόρων επιτροπών. Και ξεκινάμε με τον κύριο Μπίλτσικ της αύκο και από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως μέλη του Κοινοβουλίου εκπροσωπούμε τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και άρα για θέματα αρμοδιότητας θα πρέπει επίσης να αμφισβητήσουμε την προσωπική και πολιτική ορθότητα των μελλοντικών ε, ε, υποψηφίων επιτρόπων. Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα στα, στις παρελθούσες δράσεις του κυρίου ε, ε, Επιτρόπου και επιτρέψατε μου να τα πω όλα αυτά στα σλοβακικά. Στην η, επιστολή σας λέει ότι ένα μια ισορροπημένη επιτροπή θα χρησιμοποιήσει καλύτερα το δυναμικό. Αυτή είναι μια καλή αρχή, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Στο παρελθόν έχετε πει επανειλημμένα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρεμποδιστούν διάφορε μορφέ διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένη τη βία που, που οφείλεται στο φύλλο. Και φέτος καλωσορίσατε τη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου της Ευρώπης και Σλοβακικής Κυβέρνησης για την βία ε, των φίλων. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα απαντήσω σλοβακικά ώστε και ο, οι συμπολίτες μας στη Σλοβακία να κατανοήσουν καλύτερα ε, απευθείας μάλλον τη συνομιλία μας με τον Σολοβάκο συνάδελφο. Η ερώτηση που μου θέσατε είναι μια ερώτηση που με επηρεάζει πάρα πολύ στενά και μάλιστα διτά. Καταρχάς είμαι πατέρας δύο κοριτσιών και είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο για μένα να βλέπω πως οι κόρες μου έχουν χειρότερες προπτικές στη ζωή από ότι ο γιος μου μόνο και μόνο λόγω του ότι είναι κορίτσια. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου και όταν ήμουν υπεύθυνο για τους ανθρώπινους πόρους και αυτό επιδίωξα δηλαδή το εμείς ως ευρωπαϊκή, ε, ευρωπαϊκός διοικητικός μηχανισμός να δώσουμε το παράδειγμα. Πώς μπορούμε να θέσουμε, δώσουμε θετικά παραδείγματα ας πούμε για τη γονική άδεια. Πώς θα μπορούσαμε παρά μια σοβαρή οικονομική κρίση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θες, δώσουμε παραδείγματα όπως ας πούμε πίνακες επιδόσεων ε, ε, ε επίσης και επιδόματα για τα ζευγάρια του ίδιου φίλου. Και άλλα παραδείγματα έχουμε να δώσουμε. Ήμουν πρώτος που είπα και έθεσα φιλόδοξους στόχους για την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ψηλές και ηγετικές θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την έμφυλη βία, είμαι 100% υπέρ της κυρίας Ούρσουλα Φοντελάιεν και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε να στηρίξω τη δική της προσπάθεια, ώστε η έμφυλη βία να μπορεί να καταγραφεί ως ε, ε αδίκημα πλέον. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Μια επερώτηση έχω να κάνω. Στην δήλωση συμφερόντων σας, και στις ε, ε, παρελθούσες δραστηριότητε σας λέτε ότι ε, πρέπει να τηρούνται η ηθική και η διαφάνεια. Βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό για το χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής ώστε να υπάρχει μία σαφής πολιτική επικοινωνίας και πραγματικά με αποσυντόνισε ότι είδα ότι οι διάβλοι που έχετε χρησιμοποιήσει στην πολιτική σας εργασία στη Σλοβακία, ας πούμε, ε, δεν συνάδουν. Δεν δώσατε, ας πούμε, φέτος στη Σλοβακία καθόλου. Θα μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα δίνετε ίση πρόσβαση στα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σλοβακίας. Επιτρέψατε μου να απαντήσω στην γλώσσα μου, λέει ο Επίτροπος. Αγαπητέ συνάδελφε, πριν από λίγα λεπτά στην πρώτη σας ερώτηση, τονίσατε πόσο σημαντικό είναι να τονίσω τις αξίες τις οποίες έχω ανέκαθεν στηρίξει και εγώ τόνισα ότι στηρίζω τις ε, αξίες της Βελούδινης Επανάστασης όλη μου τη ζωή έχω στηρίξει αυτές τις αξίες και θα δείτε ότι πολλές φορές έχω αρνηθεί να ασχοληθώ με πράγματα που ήταν ενάντια. Αν έχετε τώρα κάποιες εκ των πληροφορίες ευχαρίστως να σας επικοινωνήσω, να σας διαβιβάσω μάλλον τα, τις επαφές μου με τον τύπο ε, φυσικά και έρχομαι σε επαφή με όλους όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μου. Και όχι μόνο το πράγμα αυτό, αλλά και οποτεδήποτε εμφανίζομαι δημόσια, πάντοτε περασπίζω τις ευρωπαϊκές θέσεις, γιατί... Αυτό που είναι σημαντικό για μας τους Σλοβάκους είναι να είμαστε μια ισχυρή δύναμη μέσα σε μια Ενωμένη Ευρώπη. Και το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, Τίμο Βέλκεν από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Σεύσοβιτς. Καταρχάς επιτρέψτε μου πάρα πολύ σύντομα να αρχίσω με το εξή. Με ευχαριστίες Ευχαριστώ που θέλετε να ενισχύσετε το δικαίωμα πρωτοβουλία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να είστε βέβαιο ότι θα φροντίσουμε πάρα πολύ να εφαρμοστεί. Και μια παρατήρηση για την αρχή αυτή, one in, one out. Εδώ προσκρούει σε σφοδρή απόκρουση, ε, διότι δεν είναι μαθηματικά ε, ε, ε, η ευρωπαϊκή πολιτική και ούτε κάποιο νυχτερινό μαγαζί που έχει πόρτα και ε, για να μπει ένας πρέπει να βγει κάποιος άλλος. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη διαφάνεια, διαφάνεια τους πολίτες. Αυτό το λέει και το προήμιο της συνθήκης. Αν δεν καταφέρετε να πείσετε την κυρία Φόντερ Λάιν ότι δεν χρειαζόμαστε αυτή την αρχή ένα νέο νομοθέτημα ίσον απόσυρση παλαιού, Πώς ε, θα φροντίσετε το Κοινοβούλιο και οι πολίτες να συμμετέχουν με διαφάνεια για να βλέπουν ε, ποιο νόμο καταργείται για να φέρετε ένα καινούριο. Thank you uh, this Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για σας αλλά για το ευρύτερο κοινό. Και πάλι θα ήθελα να επαναλάβω ε, την προσήλωσή μου και τη δέσμευσή μου μείωση της γραφειοκρατίας θα γίνει με κάθε αυστηρότητα αλλά και με κάθε προσοχή. Ε, και αν έχετε προτάσεις για το πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να μειώσουμε αυτό το γραφειοκρατικό άγχος, βεβαίως ε, συνομοθέτης είστε και θα σας διαβουλευθούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Πρέπει να είμαστε εταίροι και παραστάτες θα είστε στο πλευρό μας. Το, είδα και στις ε, προετοιμασ... Ε, προκαταρκτικές συνεδριάσεις που είχα στην προετοιμασία μου μαζί σας, ε, ότι έχετε πάρα πολύ καλή εμπειρία από τις τοπικές κοινωνίες. Όλη την νομοθετία λοιπόν θα, τη βλέπουμε από αυτά τα γυαλιά. Όχι απλώς να εγκρίνουμε κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη, αλλά να ανοίξουμε και το δρόμο ή τηλεοφόρο για μια Περί συλλογή ένα προβληματισμό τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι μόνο νομοθεσία, ακόμα και αν είναι σημαντική, μπορεί να δυσκολεύει τους πολίτες. Και αυτό που πραγματικά επιζητώ είναι πώς μπορούμε να κάνουμε την νομοθεσία πιο φιλική προς το χρήστη, πιο ψηφιακή. Και ίσως να διδαχθούμε και λίγο από την πληροφορική όπου εκείνοι που αναπτύσσουν τις εφαρμογές για τα κινητά μας τηλέφωνα το κάνουν ρωτώντα τους χρήστες και ακούγοντας το feedback, ε, τις απαντήσεις και όταν κάτι δεν πάει καλά, προσπαθούν να το διορθώσουν. Ε, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το ίδιο. Αν έχουμε γκρινικά που είναι πολύ βαρύ, πολύ δύσκολο ε, και έχουμε παράπονα, ας μην υποδιόμαστε ότι είναι και το απάβγασμα της ελιότητας Ας είμαστε λίγο πιο ταπεινοί και πιο ταχύ στην αντίδρασή μας, έτσι ώστε να είναι σύγχρονη η νομοθεσία μας, ενημερωμένη και όχι βαριά και φορτική. Ε, θέλετε να κάνετε συμπληρωματική ερώτηση, όχι καλύφθηκα. Ε, New Europe, με ε, Pascal Για το Renew Europe, Pascal Durand από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας κύριε Σεφτσοβίτς. Πριν από λίγο μιλήσατε για καλύτερη ενημέρωση για τα θέματα της εκπόνησης των μελετών αντικτύπου. Τώρα όμως η δημοκρατία μας αντιμετωπίζει μια νέα δυσκολία. Μένουμε σε έναν κόσμο όλο και μεγαλύτερης ε, εμπειρογνωμοσύνης και πιο λεπτομεριακό γνώσεων. Είχαμε το Dieselgate, ε, είχαμε το σκάνδαλο της γλυφοσάτης και τις μελέτες που έγιναν και την αξιολόγηση αυτού του, αυτής της δραστικής ουσίας. Και παρόλα αυτά είχαμε πολλές μελέτες περίπλοκες. Πώς όμως θα φροντίσετε ώστε οι, οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων, η καταξιδότηση πράξης, ε, και όλες αυτές οι πράξεις που ουσιαστικά εκχωρούν τη δημοκρατία στους εμπειρογνώμονες δεν θα υπόκεινται σε ιδιωτικά ή κρατικά συμφέροντα ώστε να επαναφέρουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο του όλου θέματος. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερος το γεγονός ότι δώσατε μια πολύ ζωντανή προοπτική σε όλα τα μελλοντικά μου καθήκοντα. Και πραγματικά φαίνεται πόσο είστε πριν από εμά μερικές φορές και πόσο έχει ενδιαφέρον το κοινό μας έργο και η κοινή μας προσπάθεια. Πολύ πρόοδος έχει σημειωθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά ακόμη ε, προσπαθούμε και πασχίζουμε να εφαρμόσουμε σωστά τις καταξιδότηση πράξεις και θα και να συμπεριλάβουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δώσουμε την ικανοποίηση ότι ήδη ενεργεί πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ομάδε των εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα τη καταξιδότηση πράξη, νομίζω ότι τώρα το έχουμε ε, διορθώσει και οι εμπειρογνώμονε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πλήρη πρόσβαση στα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων που συντάσσουν τις ε, μελέτες ε, αντικτύπου. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν τώρα. Άλλο για τις προπαρασκευές ομάδες εμπειρογνώμων ε, για την προετοιμασία των εφαρμοστικών πράξεων. Και εκεί καλούνται τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπειρογνώμονες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Οπότε αυτό που κατά τη γνώμη μου θα βοηθούσε πολύ στη βελτίωση της διαφάνειας είναι το εξής. Όταν μιλούμε για το ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονες που θα συμμετέχουν, να εξετάσουμε ε, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αν εκπροσωπούν ενώσει συλλόγου ή οργανώσεις, να είναι αυτές οι οργανώσεις ε, ε γεγραμμένες στο Μητρό Διαφάνειας. Επίσης, τα πορίσματα τα επιστημονικά των εμπειρογνωμόνων, ε, να είναι δημοσίως προσιτά, εκ των, εκ των προτέρων να είστε ενήμεροι για το πότε γίνονται οι συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων και να είναι πλήρης ενημέρωση. Επίσης, ε, οι εμπειρογνώμονες πληροφορικής προσπαθούν να ολοκληρώσουν αυτό το μητρό και ελπίζω του χρόνου να είναι έτοιμο και Ελπίζω το νέο εργαλείο που θα έχουμε να συμβάλλει στη διαφάνεια και να σας ικανοποιήσει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, έχω μία επερώτηση. Φυσικά, με, δια... με ιδιαίτερα αυτά που μας είπατε. Ε, ο πρόεδρος Γιουκέρ είπε, εξέφρασε την ε, ε, απογοήτευσή του, τη θλίψη του και τη μετάνοιά του ότι δεν είχε λάβει υπόψη ε, δεν είχε λάβει υπόψη του την δική μας πρόταση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. και δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μέσω τον ε, νέο οργανισμό και έναν ανεξάρτητο μέσο. Συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβα καλά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας μιλήσαμε για τα προβλήματα των εκπομπών, το διεξίδιο του άνθρακα, τα καυσαέρια. Και είπαμε κρίμα που δεν υπάρχει ανεξάρτητο οργανισμό και κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχτηκε την πρότασή μα. Τελικά είπε ότι κρίμα, είπε ο πρόεδρο Γιούγκερ, μακάρι να είχαμε έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό που θα επιφορτίζεται με τα θέματα αυτά του ελέγχου των εκπομπών. Ε, οπότε θα επανέλθει αυτό το θέμα στο πρόγραμμα εργασιών σα, ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό στην ε, στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, όντω, αυτό ήταν ένα από τα πολύ δύσκολα θέματα που ε, μας απασχόλησαν στην προηγούμενη επιτροπή. Γιατί όντω το Dieselgate, αυτό το σκάνδαλο με, με τα καυσαέρια, είχε ε, την ε, διαπλοκή που υπήρχε μεταξύ των ε, αρχών ελέγχου των κρατών μελών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και είδατε τι τραγικές διαστάσεις πήρε αυτό το θέμα και πόσο δύσκολο ήταν να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν. Και τώρα κάνουμε το πάνω δυνατό για να προλάβουμε τις νέες τάσεις όπως είναι την ηλεκτρική κινητικότητα. Και σίγουρα ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τι εκπομπέ ή για τις οδικές μεταφορές θα βοηθούσε πολύ περισσότερο και θα διευκόλυνε την κατάσταση. Το θέμα είναι η νέα επιτροπή τι προσέγγιση θα ακολουθήσει και πώς θα εφαρμόσει τις νέες προδιαγραφές που θα ε, επεξεργαστούμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Μάρκο Πίπερ από το ΕΛΚ Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς ε, ήταν ο σημαντικότερος εμπνευστή ε, για τη Συμφωνία του Παρισιού και είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τους στόχους. Δυστυχώς, κουβαλάμε πάρα πολύ γραφειοκρατική σαβούρα μαζί μας. Και ρωτώ αυτή η αρχή, one in, one out. Τι σημαίνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δέσμευση ότι θα εφαρμόσει αυτή την αρχή, ναι ή όχι. Να αποσύρεται ένας νόμος ε, για κάθε νόμο που έρχεται. Και δεύτερη ερώτηση, ε, ε, μελέτη επιπτώσεων και αντικτύπου. Ισχύει αυτό που ακούγεται και συζητείτε αυτό τον καιρό, ότι στις πρώτες 100 μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναβάλει την ε, αναθεώρηση το μελετών αντικτύπου για να φέρει όσο γίνεται περισσότερο νομοθετικό έργο. Ισχύουν αυτά που ακούγονται ή θα φροντίσετε να συνεχίζει να γίνεται καλή μελέτη επιπτώσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις χωρίς ε, ελλείμματα. Και τρίτη ερώτηση. Ωραίε και καλέ είναι αυτέ οι μελέτε αντικτύπου, αλλά στο κάτω-κάτω είναι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εσεί έχετε κάθε συμφέρον ο αντίκτυπο των δικών σα ε, ενεργειών να είναι θετικό. Έχουμε και ένα ανεξάρτητο όμω όργανο ελέγχου, ε, Regulatory Scrutiny Board. Αυτό θέλετε να το αναβαθμίσετε και να το κάνετε ε, ένα αντίστοιχο συμβούλιο ανεξάρτητο όπως υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία. Uh, Αυτή την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου. Απάντηση. Ε, το one in, one out. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι θα επικεντρωθούμε ακριβώς σαν μία ακτίνα λέιζερ ε, στο γραφειοκρατικό φόρτο που θα πρέπει ε, κάθε φορά όταν έρχεται μια νομοθεσία να αφαιρείται ε, μια άλλη ή από κάθε νέα νομοθεσία να αφαιρείται αυτό ε, το γραφειοκρατικό βάρος. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, γιατί αν το προσεγγίσει κανείς αυτόματα και μηχανικά μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη αντικτύπου και επιπτώσεων, πραγματικά χρειάζεται να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη διαφάνεια. Ξέρω ότι τώρα γίνεται συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς ε, θα μπορεί κανείς να διευρύνει τις αρχές και τους παράγοντες που θα εκτιμώνται στη μελέτη αντικτύπου. Θα ακολουθήσουμε αυτές τις συστάσεις για να γίνει ευρύτερος ο έλεγχος αυτό και στραμμένος προ το μέλλον. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου και την ανεξαρτησία της, ε, ε, θα γνωρίζετε πιστεύω ότι ε, στην τελευταία περίοδο είχαμε τρεις εξωτερικούς επιρρογνώμονες που συνεργάζονταν στην Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου και επειδή εγώ ασχολήθηκα με την Ενεργειακή Ένωση, Πραγματικά είναι πολύ αξιόλογοι αυτοί. Όταν βλέπουν ότι κάτι δεν δουλεύει καλά, δεν ε, ε, αξιολογείται σωστά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και δεν διστάζουν να μπλοκάρουν όλη τη διαδικασία και να εξασφαλίσουν ότι θα αντιστοιχεί ε, στις πολύ ψηλέ απαιτήσει για την ποιότητα της νομοθεσίας. Εγώ θέλω να τους ενισχύσω, να τους υποστηρίξω, να βελτιώσω την ποιότητά τους, να έχουν περισσότερους πόρους για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να αξιοποιούν πλήρως το κοινό ερευνητικό κέντρο για ναι, να έχουμε περισσότερα στοιχεία επιστημονικά όπου τα χρειαζόμαστε, να συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες και να είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά ό,τι κάνουμε ε, βασίζεται στην επιστήμη. Συγγνώμη, αλλά τελείωσε ο χρόνος μου. Okay. Question, Μια συμπληρωματική ερώτηση, αν επιτρέπετε. Δέκα λέει ο πρόεδρος δεν χρειαζόμαστε τρεις εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. 300 χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτά που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτη ε, επιπτώσεων και ανεξάρτητη. Είστε διατεθειμένοι να αυξήσετε και το προσωπικό. Και τελευταία ερώτηση. Είστε ε, επιτέλους υπέρ ε, ενός, ε, μιας δοκιμής υποχρεωτικής για τις μικρομεσαίες, δηλαδή αν αντέχουν οι μικρομεσαίες αυτή τη νομοθεσία. Απάντηση, ναι, ναι, το κατάλαβα, πολύ γρήγορα. Ας κοιτάξουμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε ε, την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου με τις ανεξάρτητες αρχές στα, στα κράτη-μέλη και να το συγκρίνουμε. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς στο κάτω-κάτω είναι καλή νομοθεσία, όχι βαριά και δύσκολη και προς το όφελος ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Για τις μικρομεσαίες και τη σχετική δοκιμή αυτό ήταν πάρα πολύ προσφυλές και είναι ε, στην κυρία Φόντερ Λάιεν και σε διάφορες συζητήσεις που κάναμε το ε, έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα πρέπει να τους φερόμαστε καλά γιατί πολλές φορές είναι πολύ περίπλοκη η νομοθεσία για τις μικρομεσαίες. Οπότε μάλιστα ε, θα το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό φίλτρο, ε, ένα δίκτυ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν έχετε προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, έτσι ώστε οι μικρομεσαίοι μας να μείνουν ικανοποιημένοι με τις νέες αλλαγές που θα φέρουμε. Tiene ahora la palabra Iván García del Blanco, miembro... Iván García del Blanco σοσιαλιστής από την Νομική Επιτροπή. Ah. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σεφτσοβιτς, ε, αναφέρετε προηγουμένως στην τεχνητή ε, νοημοσύνη και την ανάπτυξη της ε, της αυτής νοημοσύνης που θα σχετιστεί περισσότερο με την ψηφιακή μας ατζέντα. Εδώ τώρα οι συμπολίτε ε, υπερασπίζουν χαμηλότερη ε, νομοθετική δραστηριότητα ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Σήμερα ο κανονισμός που διέπει είναι, ε, τέτοια πράγματα είναι ο κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ε, ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία από πλευρά τη Κομισιόν θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία τη ιδιωτική ζωή και των προσωπικών στοιχείων ή μη διάκριση. Επίση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη εγγύηση του σεβασμού ε, διαφόρων ηθικών και ανθρώπινων πτυχών και να δημιουργηθεί έτσι εμπιστοσύνη στι νέε αυτέ τεχνολογίε. Πώ θα εξασφαλίσετε αυτέ οι πρωτοβουλίε υπέρ τη διευκόλυνση τη τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορου τομεί δεν θα υποσκάψει ή δεν θα υποβαθμίσει την ισχύουσα νομοθεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πώς αυτή η προστασία δεν θα είναι εις βάρος των ανταγωνιστικών πλονεκτημάτων μας. Σας ευχαριστώ κύριε Μπλάνκο για αυτή την ε, πολύ ε, διορατική ε, ερώτηση η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει και θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ εις βάθος. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή. Τι είναι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι αλγόριθμοι ή οι μηχανήματα που μπορούν ανεξάρτητα να παρατηρούν το περιβάλλον, να υιοθετούν αποφάσεις, να επικοινωνούν μεταξύ τους και μετά να ενεργούν. Και βεβαίως τέτοιου είδους ε, μηχανήματα μπορεί να υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωή, ας πούμε να δίνουν ιατρικές συνταγές, να κάνουν ιατρική εργασία, να είναι υπεύθυνοι για την αυτόνομη οδήγηση. Αγγίζει αυτό την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. Ποιος θα είναι υπεύθυνο αν κάτι πάει στραβά, ποιος ε, θα έχει στην κατοχή του τα δυτικά μας στοιχεία και ποιος θα εγγυάται τα δικαιώματά μας. Και εδώ θα πρέπει 100% να επιμείνουμε στην ευρωπαϊκή μας προσέγγιση προς τα δεδομένα και προς την ε, τεχνολογία της πληροφορίας. Άκουσα ότι οι μεγάλες εταιρείες ίντερνετ ε, στις ίπα ε, ευημερούν γιατί έχουν στην κατοχή τους το 70% των στοιχείων, των ιδιωτικών στοιχείων του αμερικανικού πληθυσμού. Στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί εμείς ε, να γνωρίζουμε ότι είναι νέο κάψιμο της οικονομίας του 21ου ε, αιώνα, αλλά ε, απ' την άλλη θέλουμε απολύτως να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά μας και να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο και ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πάντοτε αυτοί που ελέγχουν την κατάσταση. Θα είναι λοιπόν ένα από τα σοβαρά ζητήματα της Κομισιόν, πώς λοιπόν θα παραμείνουμε ε, στην πρωτοπορία, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργήσουμε με τον ευρωπαϊκό μας τρόπο. Μάλιστα, κύριε Μπλάνκο, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να προσθέσετε κάτι. Μάλιστα, παρακαλώ. Εσείς ε, απαντήσατε με πολλές ωραίες ερωτήσεις και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στα δικά μου ερωτήματα. Όμως συγκεκριμένα, πώς σκοπεύετε να έρθετε σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σε σεβασμό με τα όσα προανακοινώσατε ε, για την Ευρώπη του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για αυτή σας την ερώτηση. Όταν προετοιμαζόμουν για αυτή την ακρόαση, συζητούσα βεβαίω με του εμπειρογνώμονε για το πώ λειτουργεί το REFIT. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, μου είπαν όλοι, και λειτουργεί πολύ καλά ω πλατφόρμα. Αλλά ίσω θα πρέπει κάτι νέο να φέρουμε, μου πρότειναν οι συνεργάτε μου, κάτι το οποίο θα είναι πιο. Ε, ε, μοντέρνο, πιο σύγχρονο. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να ξυγχρονίσουμε την ομοστασία, ώστε όχι μόνο να γίνει λιγότερο φορτική, αλλά και περισσότερο προσιλωμένη στο μέλλον, να μπορεί να καλύψει αυτά που μας φέρνει ο τόσο δυναμικός αυτός τομέας. Θα δούμε λοιπόν με τους εμπειρογνώμονές μας πώς θα εξυγχρονιστούμε ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τις μελλοντικέ πλατφόρμες και όταν θα έχουμε επιτάπητο στις νέες προτάσεις θα έρθουμε εδώ στις επιτροπές σας, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω τις δικές σας συμβουλές και προτάσεις και θα ε, μπορέσουμε έτσι να οικοδομήσουμε πολιτική στήριξη για αυτή τη νέα πλατφόρμα γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε εδώ αλλά να είναι και κάτι το οποίο να αισθανθεί και ο κόσμος σεβόμαστε τις δικές τους προτάσεις. Η Μαρή από τους Πράσινους, που είναι μέρος και της Επιτροπής Ήτρε και της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ. Κύριε Σεφτσοβιτς, καλημέρα σας και ευχαριστώ που ήρθατε. Είπατε θέλετε μία ε, τεκμηριωμένη νομοθεσία. Τι γίνεται με την προστασία του περιβάλλοντος, ε, του κλίματος, της υγείας, της ε, κοινωνικής ισότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να καθοδηγούν και τις μελέτες και την ομοθεσία που στόχο έχει την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, τι γίνεται ε, με το Dieselgate και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου για τη μη δημοσίευση των μελετών για την κλειφωσάτη. Είπατε ότι θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτές οι μελέτες. Ε, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι και οι μελλοντικέ μελέτες θα είναι δημόσιες και προσιτές σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσβάσιμες και στο ευρύ κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τουσά που ήσταν πολύ ακριβής και συγκεκριμένη στην ερώτησή σας, ε, κυρίως για την υπόθεση της γλυφοσάτης. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που δεν μπορούσαν να, δεν να είχα προβλέψει ούτε καν οι συνθήκες μας τότε. Υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπουν την υποβολή προτάσεως. Ακολουθεί η συζήτηση στην επιτροπολογία. Όταν όμως δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της εξουσιοδότησης, τι γίνεται. Επίσης έχουμε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι κατά της ε, νομοθετικής πρότασης και την κοινή γνώμη στα κράτη-μέλη που είναι διχασμένη. Οπότε έχουμε εν μέρη ένα πολιτικό πρόβλημα, αλλά και πρόβλημα με την αξιολόγηση των επιστημονικών πορισμάτων και τεκμηρίων ε, των πορισμάτων που μας παρέχουν οι διάφοροι οργανισμοί μας. Και είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένω και στο μέλλον. Πάντως συμφωνώ μαζί σας ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται και να δείξουμε και στο κοινό και σε εσά που είστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών να δείξουμε ποια ήταν η επιστημονική βάση για τη συγκεκριμένη πρόταση. Και αν τα καταφέρω, ελπίζω με τη δική σας βοήθεια, να θεσπίσω αυτό το κοινό μητρό για την τεκμηρίωση και μάλιστα ένα μητρό που θα έχει διοργανικό χαρακτήρα, ε, θα φροντίσουμε ώστε όλες οι μελέτες που χρησιμοποιούνται, όλη η τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για τις μελέτες και για την υποβολή των νομοθετικών μας προτάσεων να περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αυτό διοργανικό μητρό, ώστε να είναι προσιτή η πληροφόρηση σε όλους, να μπορεί και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει την επιστημονική τεκμηρίωση που αποτέλεσε τη βάση του νομοθετικού της έργου. Έχετε επερώτηση, μάλιστα, για το θέμα της διαφάνειας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το Συμβούλιο. Η αδιαφάνεια του Συμβουλίου και η ανικανότητά του να ανταποκριθεί στις δημοκρατικές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών τροφοδοτεί αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που υποδαβλεί τη δημοκρατία και υπονομεύει την κατάσταση λόγω της αδιαφάνειας που υπάρχει. Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλλει μια, έναν απόρριτο χαρακτήρα, μια εμπιστευτικότητα και στις συζητήσεις και στα έγγραφά του. Ε, κάτι που ενοχλεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κουλτούρα του απόρριτου Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί ε, και στο Συμβούλιο μια διαφάνεια αντίστοιχη τουλάχιστον αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αν δεν τηρήσει τι συστάσει ε, τη Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια και αν τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφύγει στο δικαστήριο, θα, θα προσχωρήσετε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, αυτό, σε αυτή την προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη αδιαφάνεια του Συμβουλίου. Σα ευχαριστώ για την εύστοχη ερώτησή σα. Όντως την έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και σχετική νομολογία. Έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Δεκαπιτάνη. Πολύ σημαντική δικαστική απόφαση και μας βοηθά για το θέμα της διαφάνειας. Έχουμε αυτά τα τετράστιλα κείμενα που είναι πολύ σημαντικά και για τη διαφάνεια και για την προετοιμασία των τριμερών διαλόγων. Και γνωρίζετε, όταν ε, θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν έχει ενδιαφέρον να ε, παρουσιάσει και να ζητήσει κάποια έγγραφα, ή μάλλον ε, όταν ζητούνται κάποια έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, θα προσπαθήσω να υπενθυμίσω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ανάγκη να επανέλθει στο θέμα αυτό και να το συζητήσει με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια και με ενθάρρυνε ιδιαίτερα η Φιλανδική Προεδρία που ήδη πειραματίστηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και μιας απόπειρας να κάνει δημόσια τα έγγραφα του Συμβουλίου και ευελπιστώ ότι και οι επερχόμενες Προεδρίες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Φιλανδικής για μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Γιώχεμ Κούς από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, μέλος της Επιτροπής Γιούρη και Αύκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε, κύριε Σεφτσοβιτς. Από εδώ κοιτάξτε και λίγο δεξιά. Όταν ήρθα πριν από λίγους μήνες και ήμουν για πρώτη φορά σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή στις Βρυξέλλες, συγκλονίστηκα. Γιατί άκουσα να γίνεται λόγος για το Συμβούλιο, λες και είναι εχθρός μας. Δηλαδή το Κοινοβούλιο βλέπει ε, όχι ως αντίπαλο το Συμβούλιο καν, ως εχθρό. Και αυτό με εξέπληξε πάρα πολύ. Και στις επόμενες διεδριάσεις διαπίστωσα ότι η σχέση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο ουσιαστικά ε, φαίνεται πολύ διαταραγμένη. Για ένα τη φορά δεν έχουν δώσει απαλλαγή ε, στην οικονομική εκτέλεση του προπολογισμού του Συμβουλίου τι θα κάνετε και τι μέτρα θα λάβετε έτσι ώστε να αποκατασταθεί ή να βελτιωθεί, εν πάση περιπτώσει, η σχέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούς για την ε, απάντησή σας. Βέβαια, ε, για την ερώτησή σας, συγγνώμη, και για το όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε όσο γίνεται περισσότερο τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους όλα τα θεσμικά όργανα. Όπως γνωρίζετε, εγώ ε, θα εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι θα είμαι και συχνός προσκεκλημένος στις επιτροπές όπου σήμερα γίνεται η ακρόαση, ακόμα και στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ή όπου αλλού θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να έχετε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρειάζεται να συζητήσετε μαζί του τα θέματα συνεργασίας και τα τρέχοντα. Ε, εξίσου θα εκπροσωπώ την Κομισιόν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο προετοιμάζει τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Κορυφής και ασχολείται με εγκάρσια θέματα όπως το πολιετές δημοσιονομικό, όπως ε, η πολιτική συνοχή, η διεύρυνση και άλλα τόσο σημαντικά για σας. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα μεταξύ των συνομοθετών, Συμβουλίου και ε, Κοινοβουλίου, να είναι όσο γίνεται πιο αγαστή. Και έτσι ε, προσεγγίζουμε και τους τριμερείς διαλόγους, όπου επενδύουμε τεράστια ενέργεια για να ε, εξασφαλίσουμε ότι οι θέσεις συμπλησιάζουν όσο μπορούν πριν την τελική διαπραγμάτευση για να έχουμε κάποιες λογικές προοπτικές επιτυχίας. και σύμφωνα και με τη συμβολή ε, του εκπροσώπου ε, της Γενικής Γραμματείας λέει θα πρέπει να τηρώ τις ίσες αποστάσεις. Δηλαδή ε, η έκφρασή του είναι να είμαι εξίσου μακριά. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Θέλω να πω ότι θέλω να είμαι εξίσου κοντά γιατί καμιά φορά θέλω να μεταφράζω τα παράπονα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να ε, εξηγώ τη θέση του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο για να βρίσκουμε μια λύση, όπως κάναμε και με διάφορες διοργανικές συμφωνίες ε, που είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε όπως όταν ήμουν για πρώτη φορά επίτροπος. Ο κύριος Κούς, έχω καλυφθεί, ευχαριστώ, δεν έχω συμπληρωματική ερώτηση. E e και τώρα ο κύριος Ζαμπάσκι, Πολύ δραστήριο σήμερα ο κύριος Ζαμπάσκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεύτσοβιτς, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, οι διαθεσμικές σχέσεις πολλές φορές υποφέρουν από διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Αυτό ε, ισχύει ας πούμε έναντι των ε, ανατολικών ευρωπαϊκών κρατών. Ας πούμε το, η για την κινητικότητα. Κάνουμε λόγο για πράσινη ενέργεια. Όμως σε αυτό το, το, τη δέσμη κινητικότητας προβλέπεται ότι άδεια φορτηγά επιστρέφουν, ε, διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα εκπέμποντας διοξίδιο του άνθρακα μόνο και μόνο ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δυτικών εταιριών. Και αυτό βεβαίως ε, τοποθετεί τις ε, αεροτολικές εταιρείες σε μειονεκτική θέση. Αυτή είναι μια αντίθεση βέβαια. Ε, μιλάμε για ενέργεια, για πράσινη ενέργεια και για μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όμως πώς θα λύσετε αυτό το συγκεκριμένο επίμαχο ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την ερώτηση και θα πρέπει να πω πως προς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 απογοήτευση του Επιτρόπου Μεταφορών του και Μπούλτς, της κυρίας Μπούλτς και εμένα είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα κρεμεί. Και αυτό γιατί δεν καταφέραμε να φτάσουμε, να βρούμε μάλλον την συντριπτική συνένεση που θα κάλυπτε την πλειοψηφία των 100 μελών και των μελών του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ξέρετε ότι ε, αυτό που συζητήσαμε ήταν πόσες μέρες θα, θα έχουν μάλλον μάλλον οι οδηγοί των φορτηγών για τις διεθνείς μεταφορές, πόσες μέρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το καμποτάζ, ποιοι είναι οι κανόνες για την ε, ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία ανάπαυση και ούτω καθεξής. Ε, Νομίζω πως τελικά ε, μπήκαμε σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες, πράγμα που κατέστησε την λύση εξαιρετικά περίπλοκη. Νομίζω πως κατά κάποιο τρόπο χάσαμε ε, την αρχική ιδέα, τον αρχικό στόχο αυτής της πρότασης που ήταν το να μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε αυτές τις εταιρείε ε, τις εικονικές εταιρείε που και να αποφύγουμε και περιπτώσεις όπου ε, εταιρείες ε, πολύ κακόφημες εκμεταλλεύονται τους ε, οδηγούς και τους κάνουν να διαφωνούν μεταξύ τους και έτσι τους εκμεταλλεύονται, τους τρέχουν τους μένα αντίον των δε. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε με αυτή την κατάσταση γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να εξασφαλίσουμε πως ε, οι οδικές μας μεταφορές θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές, πως θα μπορέσουμε καλύτερα να τις συνδυάσουμε με τους σιδηροδρόμους, να χρησιμοποιήσουμε ε, καλύτερα τα φορτηγά μας, να μην μένουν χωρίς φορτία. Ε, ναι, αλλά μιλήσαμε για διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Μια μεγάλη γερμανική εταιρεία ε, προγραμματίζει να μεταφέρει την παραγωγή της στην Τουρκία. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια συμφωνία για το επίπεδο της κρατικής ενίσχυσης Εκπρόσωποι αυτής της εταιρεία λένε ότι πηγαίνουν στην Τουρκία διότι μπορούν να παρακάμψουν ε, τους κανόνες περί επιδοτήσεων. Ε, στην Τουρκία δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, αλλά ούτε και οικολογικές προδιαγραφές, για να μην μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές ε, διαδικασίες. Τι θα κάνει λοιπόν η Κομισιόν αυτή, η γερμανική εταιρεία δεν είναι ιδιωτική εταιρεία, συμμετέχει ο Πρωθυπουργός της Εξονίας στην εταιρεία αυτή. For, for, uh, this question. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, δεν έχω ε, ενδελεχείς πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά θα σας απαντήσω πιο γενικά, πιο διαρθρωτικά. Το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων ε, τρίτων χωρών προς επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στις εισαγωγές ε, προϊόντων από τρίτες χώρες που έχουν ε, μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα από το δικό μας, από την ευρωπαϊκή παραγωγή δηλαδή. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί και να δείξουμε μεγαλύτερο στένος στις εμπορικές μας σχέσεις με τις τρίτες χώρες και να σταματήσουμε πρακτικές όπου ουσιαστικά ε, Παρατηρούμε τις εταιρείε μας ε, να έχουν φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή και μεταπίεση και μετά ε, εισάγουμε ε, ρηπογόνα εντό εισαγωγικών προϊόντα από χώρε με χαμηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε έναν φόρο προσαρμογή στον άνθρακα στα σύνορα για να εξισώσουμε τις ηθίκες ανταγωνισμού εντός και εκτό της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα από τρίτες χώρες που δεν ε, εστερνίζονται την ανάγκη μας να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές. Ο κύριος Γιάρα από το ΕΛΚ, της Επιτροπής Μεταφορών. Αναφορών, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, από την Επιτροπή Αναφορών έχω αναλάβει να σας ρωτήσω. Παίρνουμε πολλές αναφορές για περιβαλλοντικά θέματα ρήπανση περιβάλλοντος και έργα που απειλούν το περιβάλλον. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν είναι ακόμα στο στάδιο του προγραμματισμού, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε πεπισμένοι ότι τα κράτη-μέλη σέβονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο σύνολό της. Αν έχει περάσει η φάση του σχεδιασμού, φτιάχνουν γρήγορα τα έργα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα μπορεί να φτιάξεις ένα πάρκο ψυχαγωγίας διασκέδασης, ένα φυσικό δρυμό. Και ε, μετά δεν βοηθούν οι διαδικασίες παραπομπής ε, επί παραβάση στο δικαστήριο των κρατών. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως, στα πρώιμα στάδια και όχι όταν έχουν κατασκευαστεί τα έργα. Μπορείτε δηλαδή να σκεφτείτε ότι θα προσφεύγετε στο δικαστήριο ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού ενός έργου. Ε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας κύριε Γιά. Να πω μερικά ε, ε, πράγματα έτσι, διαρθρωτικά. Εγώ θέλω να έχουμε σχέση υψηλής ποιότητας με την Επιτροπή Αναφορών, γιατί κατανοώ πόσο μεγάλη είναι η ματέωση και για σας και για τον αναφέροντα όταν δεν παίρνουν ε, μια απάντηση εγκαίρωση, παίρνουν μια τελείως γραφειοκρατική και καθόλου ικανοποιητική απάντηση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να εργαζόμαστε με τρόπο πολύ ειλικρινή και να λέμε από την αρχή για κάποιες αναφορές ότι δεν εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα και ψάξτε τον αρμόδιο. Σε εκείνα όμως που εμπίπτουν στη δική μας θα πρέπει να είμαστε πιο στεναροί. Και ε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν έχουμε ε, τέτοια προβλήματα γύρω από περιβαλλοντικές άδειες ή περιβαλλοντικές μελέτες. Πολύ συχνά γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές αναφορές που έχουν να κάνουν με αεροπορικές εταιρείες και πώς φέρονται στους επιβάτες, στους πελάτες τους. Ας έχουμε λοιπόν μια διαρθρωτική συζήτηση στην Επιτροπή σας για αυτά τα θέματα ο Επίτροπος, οι υπηρεσίε του να σας απαντούν σωστά και να απαντάτε στους πολίτες για να το βλέπουμε σοβαρά για τις ε, μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου στην Ευρώπη κάθε χρόνο και δεν υπερβάλλω. Μπορεί να έχουμε δεκάδες χιλιάδες ε, μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου που γίνονται σε επίπεδο κρατικό, περιφερειακό, ακόμα και δήμου. Εκεί θα πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο τρόπο να αντιμετωπίζουμε ε, τα θέματα αυτά που μας αφορούν. Δεν έχει νόημα μεγάλο να μπαίνουμε σε συζητήσεις με ένα κράτος μέλος όταν έχει τελειώσει ήδη ένα έργο, ένα κτίριο. Uh, uh, ε, ε, αλλά πώς θα εστιάσουμε ε, όταν δούμε ότι κάτι έχει πάει στραβά να επέμβουμε και να συνεργαστούμε. Στο σκεφτούμε αυτό πώς θα γίνει η συνεργασία στην Επιτροπή Αναφορών και πώς θα το καταφέρουμε με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Συμπροματική ερώτηση του κύριου Γιάρ. Επιτρέψτε μου μια επερώτηση. Η Επιτροπή Αναφορών βασίζεται στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα πρέπει να έρχεται το αργότερο τρεις μήνες ε, από την ημερομηνία ε, που έχει ζητηθεί η απάντηση. Θα βοηθήσετε να εγγυηθείτε ότι θα τηρείτε αυτό το τρίμηνο ουσιαστικά γιατί ε, συχνά έρχεται η απάντηση καθυστερημένα και φτάνει και σε μας. Μπορούμε να κλείσουμε μια μεγάλη συμφωνία, ένα deal ότι θα τηρήσετε το τρίμηνο. Θα ήταν μια πολύ καλή αρχή αυτή. Κύριε Γιάρα, ναι, να κάνουμε αυτό το deal, αυτή τη συμφωνία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας απαντώ εντός του τριμήνου. Αν με βοηθήσετε κι εσείς να ξεκαθαρίσουμε όλα τα θέματα τα οποία δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι και το ξέρετε κι εσείς κι εμείς αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό και να μας στέλνετε πραγματικά μόνο τις αναφορές για τις οποίες μπορούμε να κάνουμε κάτι και είμαστε αρμόδιοι, θα κάνω ό,τι μπορώ να σας έχω μια καλή απάντηση εντός του τριμήνου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας πάντα για να έρχεται στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινοί και απέναντι στους πολίτες. Μην φέρνουν αναφορές που δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και το γνωρίζουμε, να το λέμε αμέσως, για να μην απογοητεύονται οι άνθρωποι και να τους ταλαιπωρούμε, να κρατάμε ανοιχτή την αναφορά και μετά να πούμε «Α, κοιτάξτε, την είδαμε, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα, ε, ξαναγυρίστε στο εθνικό επίπεδο». Ε, αν γίνει αυτό, με πολύ μεγάλη χαρά να το κάνω και προβλέπω στη συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Από το Renew ε, το λόγο έχει ε, η Ευρωβουλευτής Σράινμαχερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τους σωρευτές που αναφέρετε στην επιστολή της αποστολής σας. Πώς θα φροντίσουμε ώστε να είμαστε στην πρωτοκαθεδρία της ανάπτυξης και παραγωγής της τεχνολογίας του μέλλοντος, γιατί θεσπίστηκε αυτή η συμμαχία για τους ορευτέ, Εσείς εξασφαλίσετε το συντονισμό του έργου της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι μελλοντικέ τεχνολογίες. Οπότε πώ θα σχηματίσουμε τι απαραίτητες συμμαχίε, ώστε όντως να έχουμε καινοτόμες τεχνολογίες και να τις παράγουμε εμείς ίδιοι στην Ευρώπη αντί να τις εισάγουμε. Δεν, έχω, δεν θα πρέπει να περιμένουμε άλλα μια πενταετία για την επόμενη συμμαχία, μετά τη συμμαχία των συσσωρευτών. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις καινοτόμες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της νεοτεριστικής μας βιομηχανίας και να τις αξιοποιήσουμε. Πώς λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική πρόβλεψη και διορατικότητα ώστε να κρατήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να πω δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τους Ισορρευτές και θα τη συνδέσω με άλλου τομείς στρατηγική. Στη Συμμαχία για τους Ισορρευτές το πιο δύσκολο τμήμα ήταν ε, η έναρξη. Γιατί έπρεπε να πείσουμε τους πρωτοπόρους της βιομηχανίας ότι η να αφήσουμε το παρελθόν ε, και τον ντίζελ και να επικεντρωθούμε στις ισορρευτές και το υδρογόνο που είναι οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Επίσης, ε, οι ισορρευτές δεν είναι ένα απλό προϊόν. Έπρεπε να τους πείσουμε ότι είναι στρατηγικό στοιχείο των μελλοντικών ε, οχημάτων. Και το λογισμικό και οι ισορρευτές είναι το 80% της αξίας του οχήματος και Σίγουρα οι άλλοι δεν θέλουν να εξάγουν μπαταρίες μόνο στην Ευρώπη, στι αλλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, και σίγουρα στο μέλλον πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά οχήματα θα είναι ηλεκτρικά. Και αν είναι να το αγοράζουμε made in China, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Και αν δεν θέλουμε τα μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα να είναι κινέζικα, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ε, βιομηχανία μας και ίσως ε, θα πρέπει να περάσουν ακόμη δύο χρόνια για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να παράγουμε συσσωρευτέ που θα είναι καλύτερης ποιότητα από του ασιατικού, πιο φιλοπεριβαλλοντικοί, με προηγμένο λογισμικό και ταυτόχρονα να επενδύσουμε στην επόμενη γενιά των συσσωρευτών, ώστε όταν περάσουμε στην τεχνολογία της ε, στερεά, μπαταρίας, του σωρευτής στερεάς βάσης, να είμαστε έτοιμοι για να αισθανιστούμε τη νέα τεχνολογία. Οπότε θα πρέπει η βιομηχανία, οι ηθήνοντες πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ε, και τα χρηματοδοτικά μέσα και οι μηχανισμοί να συμβάλλουν ώστε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις καινοτόμες επιχειρήσεις και να επεκταθούμε και σε άλλους στρατηγικούς τομείς. Γι' αυτό θα ήθελα αυτές τις ευθύνε που έχω, τις αρμοδιότητες περί πρόβλεψης, να τις αξιοποιήσω και στο τομέα αυτό, ώστε να έχουμε πραγματικά βιομηχανικά σύμφωνα, ώστε να διασφαλίσουμε το μέλλον μας ε, στην πρωτοκαθεδρία του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Έχετε περώτηση? Μάλιστα. Στην προεκλογική εκστρατεία εν των ευρωεκλογών, κάτι που άκουγα συχνά από του ψηφοφόρου είναι οι Βρυξέλλε είναι πολύ μακριά, θεσπίζουν ε, περιττέ νομοθετικέ διατάξει. Εσεί μιλήσατε για την αρχή ένα μπαίνει, ένα βγαίνει, one in, one out και την ε, ελάφρυση της ε, υπερβολικής κανονιστικής επιβάρυνσης. Πώς όμως θα εμπλέξουμε σε αυτό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δούμε τι ακριβώς χρειάζονται και πώς επηρεάζονται από το ενωσιακό δίκαιο. Φυσικά, φυσικά και θα το κάνω. Και όσο ήμουν στις Βρυξέλλες ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα για τον κοινωνικό διάλογο και είδα πόσο χρήσιμο θα είναι ε, και πώς θα είναι χρήσιμη νέα προσέγγιση στις περιφέρειες που εξαρτώνται από τον άνθρακα και ε, κάνουν τη μετάβαση προς μια διαφορετική οικονομία. Και είναι θέμα ε, που σχετίζεται με τις μεταφορές, αλλά σίγουρα οι κοινωνικοί εταίροι ενδιαφέρονται για τις διαβουλεύσεις. Και στις ε, σχετικές διαβουλεύσεις που θα έχω θα υπάρχουν και εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φυσικά. Πάντως Έλαβα το μήνυμά σας και αν όντω πρέπει να εξετάσουμε το διοικητικό άχθο, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έξυπνοι και να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία που έχουμε, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα ψηφιακά μέσα και να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε το διοικητικό φόρτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε οποιαδήποτε σχόλιο ή feedback από εσά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι χρήσιμο. Και μας ενδιαφέρει να είμαστε απτοί και συγκεκριμένοι, να ρωτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ποια συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, ποιο νομοθετικό μέτρο σας κάνει τη ζωή δύσκολη. Να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να ξέρουμε ακριβώς τι προβληματίζει και τι επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Αυτό θα, είναι, θα μας εξασφαλίσει και πιο αποτελεσματική δράση. Ευχαριστώ. Next question is from Mr. Castaldo, from the non-aligned group and from the Af Ο κύριος Καστάλντο, μία γεγραμμένος από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, μεγάλη χαρά μας που είστε σήμερα εδώ για αυτήν την αντιπαράθεση. Η δράση των θεσμών και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να βασίζονται στη συμμετοχική δημοκρατία, ε, να εγγυώνται τις αρχές της διαφάνειας, της ε, κοινή διάδοσης και γρήγορη διάδοσης της πληροφορίας στους πολίτες. Άκουσα τα όσα είπατε όσον αφορά τον σεβασμό της απόφασης δεκαπιτά κάνει από τις ε, νομολογίες. Δηλαδή θα ήθελα επίσης να μιλήσω με βάση τα όσα είπατε και σε κάποια από τι γραπτές σας απαντήσεις. Όταν είπατε πως είστε δεσμευμένο, να γίνονται οι διαπραγματεύσει ε, και με βάση το κοινό μητρό διαφάνεια. Αυτό ε, θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν αν κατά τη γνώμη σα, μάλλον πώ σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τι διαπραγματεύσει εφόσον το Συμβούλιο έχει πρόθεση να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα μπορούσε άμεσα να διβελτιώσει άμεσα τη διαφάνεια και την ε, δημοκρατική διαδικασία και αυτό ε, μάλιστα ταχύτητα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καστάλτο. Όσον αφορά το Μητρό Διαφάνειας, θυμάμαι πως ξεκινήσαμε με την ανανέωση του συστήματος που είχαμε τότε και νομίζω πως ήταν περίπου 8-9 χρόνια πριν έπρεπε να προσαρμόσουμε αυτό το μητρό στις διάφορες εταιρείες, συνδέσμους, μικιό, ε, ε, όλους τους τομείς της ζωής δηλαδή και όλους όσους ήθελαν να είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής συζήτησης και της ευρωπαϊκής νομοθετικής συζήτησης και νομίζω πως αυτό το καταφέραμε και σήμερα νομίζω πως το Μητρό Διαφάνειας είναι πραγματικά σημείο αναφοράς εάν συγκρίνουμε οποιαδήποτε χώρα στην Ένωση ή στον ΟΣΑ ή και τη ΣΥΠΑ αν συγκρίνουμε. Ε, υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα όπου θα πρέπει να συνεχίσουμε να, τη συζήτησή μας και πιστεύω πως και εδώ είναι ε, κάτι που εκκρεμεί από την τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Πώς μπορούμε αυτό το μητρό της διαφάνειας να το κάνουμε ακόμα πιο δημοφιλές για το Ευρωκοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Ξέρω πως αυτά τα ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητα. Πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία και ε, για μας και για σας, γιατί είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, ε, είστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών ε, ε, πρέπει να λογοδοτήσετε και πρέπει να εξασφαλίσουμε πως το σύστημα της διαφάνειας ε, θα λειτουργεί εύρυθμα. Το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο και νομίζω πως αν καταφέρουμε όλοι οι τρεις θεσμοί να έχουν την ίδια προσέγγιση στο Μητρό Διαφάνεια θα εξυπηρετήσουμε πραγματικά τους Ευρωπαίους πολίτες και θα δώσουμε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλες τις δημοκρατίες αυτού του πλανήτη για το πώς με διαφάνεια ε, εμεί αντιμετωπίζουμε τους εκπροσώπους των ε, εταιριών ε, ή των διαφόρων μάλλον συμφερόντων όταν έρχονται να συνομιλήσουν μαζί μας. Και Συγγνώμη που παρασύρθηκα με το Μητρό Διαφάνειας και δεν είχα χρόνο ε, να απαντήσω στην ερώτηση για την απόφαση του καπιτάνη. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, αν γίνει επερώτηση να απαντήσω στη συνέχεια. Μάλιστα, θέλετε να κάνετε περώτηση. Ναι, σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας ε, και θα ήθελα επίσης να καταλάβω αν όντω θα έχετε την πρόθεση να υποβάλλετε νομοθετική πρόταση για, για, για, για κανονισμό για να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Και έπειτα θα ήθελα να δω, να καταλάβω ε, πώς θα μπορέσετε να προωθήσετε τα θέματα τα πολύ σοβαρά σε άλλους τομείς. Ε, το Συμβούλιο ξέρω πως ε, και εδώ για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό και θέλω να καταλάβω πώς σκοπεύετε εσείς να ε, δράσετε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα έρευνας. Εάν ως Κοινοβούλιο θέλουμε ας πούμε να φέρουμε ένα θέμα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ποια θα ήταν η θέση σας, πώς θα βλέπατε εσείς μια τέτοια θέση και θα ήσασταν έτοιμος ίσως και να τη στηρίξετε. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω την πρώτη σας ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το Μητρό Διαφάνειας, αυτό που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση, η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Να δούμε πώς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι τμήμα αυτής της διαδικασίας και είμαι απόλυτα πρόθυμος για κάτι τέτοιο να το συζητήσουμε αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα έρευνας, είναι κρίμα που από το 2012 έχει κολλήσει το θέμα. Έχετε απόλυτο δικαίωμα να ζητάτε αλλαγή της παροχημένης ε, νομοθεσίας για το θέμα αυτό και αντιλαμβάνομαι, είναι ευνόητο ότι θέλετε τις απαραίτητες αρμοδιότητες και εξουσίες ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την έρευνα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική μου πρόταση είναι η εξή. Θα οργανώσω μία συνάντηση με την παρούσα και τις μελλοντικέ προεδρίες και μπορούμε να έχουμε συζήτηση και με τους συντονιστέ των επιτροπών μας για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ή μήπως έχουμε τόσο γεφύρωτες διαφορές που θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη μια πενταετία από την υποβολή της πρότασης ή μήπως μπορούμε να αναζητήσουμε μια επικοδομητική συμβαστική λύση ώστε να σας κατοχυρωθεί το δικαίωμα έρευνα που εύλογα το διεκδικείτε και ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη κάποιοι νομικοί περιορισμοί που ε, μας που υποβάλλουν κυρίως οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και τους επισημαίνουν. Ο κύριος Πιζάπη έχει το λόγο τώρα που σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι μέλος Επιτροπής ε, ΑΦΚΟ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις γραπτές σας απαντήσεις και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις που δώσατε μέχρι τώρα. Έχει προφανώς αναδειχθεί ε, ότι η προτεραιότητα αυτής της θητείας θα είναι να βρεθούν οι τρόποι για να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό που προσφέρουν οι συνθήκες ώστε να βελτιωθούν ε, και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η υποψήφια πρόεδρος στηρίζει και το είπε μάλιστα στη διάρκεια μιας ε, ολομέλειας στο Στρασβούργο ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατάργηση της ομοφωνίας για τα πολιτικές που αφορούν το κλίμα, την ενέργεια, τις κοινωνικές υποθέσεις και την φορολογία. Εγώ σας ρωτώ, συμμερίζεστε αυτή τη στιγμή πριν να μπορέσετε να αλλάξετε και να μιλήσετε για αυτή την ισότητα που δεν, ισχύει, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εσείς συμφωνείτε να περάσουμε από τις ειδικέ στις ε, απλές διαδικασίες, δηλαδή στην ειδική πλειοψηφία αντί για ομοφωνία και σε ποιους τομείς θα στηρίζετε την εφαρμογή των ρητρών πασαρέλας ε, σε, σε, για, την γενική νομοθεσία όσο και για την τομεακή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πισάπια για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα όντως θα απασχολήσει την ε, ε, Επιτροπή μας. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε μια γεωπολιτική επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεσότερη δράση. Και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, που για πολλούς και διάφορους λόγους ένα ή δύο κράτη μπορούν να οδηγήσουν σε παράλυση της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να οδηγήσουν σε διέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν σταδιακά να περάσουμε από τον κανόνα της ομοφωνίας στον κανόνα της ενισχυμένης πλειοψηφίας, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά πιο ευέλικτη και μπορεί να υιοθετήσει πιο γρήγορα τις αποφάσεις της. Αυτό το έθεσε και ο συνάδελφος Μπορέλ. Ε, σίγουρα η επικοδομητική αποχή θα μπορούσε να είναι λύση σε τομείς που θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Βέβαια, οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διαπιστώσατε και από το σχέδιο για τις πρώτες εκατομέρες, αφορούν κυρίως τα κοινωνικά θέματα. Κατώτατος μισθός, διαφάνεια των αμοιβών, το Green Deal, περιβαλλοντική συμφωνία και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας για τις πρώτες 100 και φυσικά η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Νομίζω ότι όλοι θα υποφεληθούμε αν περάσουμε στους τομείς αυτούς σταδιακά από την ομοφωνία στην ενισχυμένη πλειοψηφία. Όπως ξέρετε ήμουν αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση στην προηγούμενη Επιτροπή και θα ήταν πολύ ευκολότερα τα θέματα της ε, φορολογίας, της ενέργειας ε, ε, υπόκειντο στην αρχή της ενισχυμένης πλειοψηφίας και όχι της ομοφωνίας. Για μερικές χώρες όμως βέβαια η θέσπιση του φορολογικού συντελεστή είναι ιερό και απαραβίαστο ζήτημα και άπτεται της εθνικής κυριαρχίας, οπότε θέλουν ομοφωνία. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι φόρους θα μπορέσουμε να εισπράξουμε και να επιβάλλουμε χάρη σε μια πιο ευέλικτη και ελαστική διαδικασία ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Κύριε Πιζάπια, θέλετε ερώτηση. Μάλιστα σύντομα. Είμαι ευχαριστημένος από την απάντησή σας που με πείθη και γιατί ο, ο κίνδυνος μιας τέτοιας ακρόσης είναι να τα γενικεύσουμε όλα και να μην απαντήσουμε σε τίποτα συγκεκριμένα. Ενώ εσείς εδώ συγκεκριμενο... συγκεκριμενοποιήσατε την απάντησή σας. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πλανήτη μας και για το μέλλον της Ευρώπης. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το όσα κάνατε αυτά τα τελευταία χρόνια για την Ευρώπη, αυτά που κάνετε ακόμη ως ε, ε, τμήμα της ε, σημερινής Κομισιόν και είμαι βέβαιος και ότι στο μέλλον θα κάνουμε μαζί και άλλα περισσότερα. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Πιζάπε για τα ε, καλά του λόγια και εκτιμώ πολύ την υποστήριξη που έχω από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Τι κάναμε για την Ενεργειακή Ένωση, ιδιαίτερα για την μετρίαση των κλιματικών αλλαγών, το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Συμφωνίας του Παρισιού και η υποστήριξη μάλλον της Συμφωνίας του Παρισιού στη Νέα Υόρκη ήταν μια από τις πιο περήφανες στιγμές της διαδρομίας μου και ξέρω πως πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξή τους. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια ακόμα μια φορά. Ε, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Σάγερ, ε, ευχαριστώ κύριε υποψήφιε πρόεδρε. Ένα από τα πιο καυτά θέματα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τις συντρέχουσες αρμοδιότητες. Τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σιγά σιγά ροκανίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και τις ε, ε, οικειοποιείται και τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι δεν έχουν ε, δυνατότητα αντίδρασης. Άκουσα στις απαντήσεις σας, πολύ είπαν ναι, ότι ε, όταν, και όταν δεν είστε βέβαιοι για τις νομοθεσίες και για τις προτάσεις δεν θα τις υποβάλλετε. Όταν ε, όμως ε, κινήθηκε η διαδικασία κίτρινης κάρτας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα απέρριψε όλα λίβδιν. Ορισμένοι αυτό το θεώρησαν αλαζονία και υπεροψία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα ε, λαμβάνει περισσότερο υπόψη ε, τα διάφορα κοινοβούλια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μόνο ε, ε, σε μία από τις τρεις περιπτώσεις η διαδικασία κίτρινης κάρτας ε, ευωδόθηκε. Ευχαριστώ κύριε Σάγερ για την ερώτηση αυτή. Νομίζω η καλύτερη απάντηση, η καλύτερη προσέγγιση είναι να έχουμε μια πιο πολιτική στάση και να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη διαδικασία κίτρινης κάρτας. Πιστεύω σήμερα ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαμαρτύρονται. Θεωρούν ότι 8 εβδομάδες είναι πολύ ε, σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα πρέπει σε αυτό το δίμηνο να συνυπολογίζονται περίοδοι διακοπών, όπως είναι η περίοδοι του, τέλους του έτους, α πούμε, όταν είναι κλειστά τα κοινοβούλια, ε, θα πρέπει να είμαστε πιο προδραστικοί στην προετοιμασία ε, συνολικών απαντήσεων, ολοκληρωμένων, όχι τυπικών γραφειοκρατικών σε κάθε κοινοβούλιο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια προβλήματα και έρχονται ε, να απευθυνθούν σε εμά με τα ίδια θέματα, ας είμαστε λίγο πιο πολιτικοί και να προετοιμάζουμε μια απάντηση που να απαντά ουσιαστικά στο θέμα που θέτουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ελπίζω αυτό να ε, μπορούσε να λύσει κάποια από τα προβλήματα. Και κάτι άλλο σημαντικό είναι να προσκαλούμε στις Βρυξέλλες πιο συχνά εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για να συζητούν με τους ομολόγους τους Ευρωβουλευτές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εμείς όσο γίνεται περισσότερο, όσο πιο συχνά μπορούμε να πηγαίνουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια για να συζητούμε θέματα που τους απασχολούν. Ελπίζω να μπορέσετε να επιφεληθείτε περισσότερο από την έκθεση που έκανε η ειδική ομάδα που συστάθηκε από τον πρόεδρο και πιστεύω ότι η αρχή της ενεργούς επικουρικότητας, δηλαδή σε συντονισμό εκ των προτέρων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα βοηθήσει να ε, διασκεδαστεί αυτή η αίσθηση που έχουν ότι δεν τους παίρνουμε αρκετά στα σοβαρά. Ε, έχετε δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ πολύ σύντομος να είστε. Ναι, ο κύριος Σάγερ, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Μου αρέσει. Αλλά πρέπει να πω ότι πολλές φορές Υπάρχουν θέματα προστασίας των μειονοτήτων. Ε, και εσείς, όπως και εγώ, προερχόμαστε από την Κεντρική Ευρώπη. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, υπάρχουν διαφορετικοί αντίκτυποι ε, και επιπτώσεις ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Προηγουμένως κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν το θέμα της κινητικότητας ή η εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνησαν διαδικασία κίτρινης κάρτας κάποια εθνικά κοινοβούλια. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι είναι διαφορετικές επιπτώσεις των ίδιων νομοθετημάτων στα διάφορα κράτη-μέλη, αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ υπόψη μας. Ναι, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαίωμα πρωτοβουλία, αλλά ακριβώ γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα σκέφτεται αυτά πριν κάνει νομοθετικέ προτάσει για να αποφεύγονται τέτοιε κίτρινε κάρτε ή κόκκινε. Ε, τηλεγραφικά να απαντήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο δημόσια και ιδιωτικά η εκλεγμένη πρόεδρος ε, τι θα κάνει με αυτά τα θέματα θα πρέπει αυτές οι εντάσεις και τα, ε, ε, τα χάσματα Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος να ε, καλυφθούν. Πολύ σοβαρά το παίρνει αυτό υπόψη της και θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι ενωμένη αλλά και να αισθάνεται ενωμένη και πάλι. Και είναι πολύ δύσκολο πιστεύω σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσεις κάτι ε, έτσι να επιβάλλεις κάτι ε, όταν ανθίστανται στεναρά κάποια κράτη-μέλη, ακόμα και αν είναι μειονότητα αυτή. Θα πρέπει πάντα να συζητούμε, να διαπραγματευόμαστε ξανά και ξανά και να αναζητούμε τις καλύτερες λύσεις για όλους. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια λύση βιώσιμη με υποστήριξη από όλους που θα ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Μανώ Μπρή έχει το λόγο από την ΚΟΕ. Είναι μέλος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Καλημέρα σας. Βρίσκομαι στα αριστερά σας. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα που δεν ακούσαμε μέχρι στιγμή στην ακρόαση. Παρόλο που είναι πολύ επίκαιρο και ενώ την εξέταση από το Κοινοβούλιο και την Νομική Επιτροπή την σύγκρουση συμφερόντων των υποψηφίων, κάποιων υποψηφίων επιτρόπων. Γνωρίζετε ότι για δύο επιτρόπους κρίναμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Άρα δεν είναι σε θέση, κατά τη γνώμη μας, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Εσείς μιλήσατε για ένα ισχυρό κοινοβούλιο, για ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχική σας δήλωση και σας ευχαριστώ. Αυτό που συγκράτησα όμως από την όλη διαδικασία ήταν, ήταν ταραχώδης, χαοτική και δεν νομίζω να έχει κανείς διαφορετική άποψη από την ομίγυρη. Και επίσης ε, η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από ε, φανείς δυσκολίες, περιορισμένη πρόσβαση πληροφορίες, μέσα εξακρίβωσης της ακρίβειάς τους και μια διαδικασία γενικώ που μένει σε μεγάλο βαθμό πολιτική. Κάτι που ε, πλήττει ακόμη περισσότερο και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς ως πρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις, τι προτείνετε για να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη μας στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτίθεστε να συστήσετε μια πραγματικά ανεξάρτητη επιτροπή, ανεξάρτητο φορέα ε, ε, μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου που θα έχει και τα μέσα και το χρόνο και τις αρμοδιότητες να ελέγχει τους υποψηφίους επιτρόπους πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να απαντήσω στα αγγλικά γιατί είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα, πολύ λεπτό και ε, αρκετά νομικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο για μένα να σχολιάσω ένα τόσο πρόσφατο θέμα, μια τόσο φρέσκια κατάσταση που αφορά δύο υποψηφίους επιτρόπους, δύο συναδέλφους μου. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το θέμα είναι της αρμοδιότητας Επιτροπής Γιούρη και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, της εκλεγμένης Πρόεδρου. Πάντως συμφωνώ μαζί σας ότι από τη νέα κατάσταση είναι σαφές ότι η Επιτροπή Γιούρη σωστά προσπάθησε να διαλευκάνει την, το θέμα της σύγκρουση φερόντων και ασχολήθηκε πολύ διεξοδικά και περιστατωμένα και σωστά έπραξε με το ζήτημα αυτό. Και το δεύτερο σκέλος ερώτησής σας είναι πολύ εύστοχο, γιατί θυμάμαι όταν συζητούσαμε τον εξυγχρονισμό του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και τότε για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε και το διοντολογικό κώδικα για τους επιτρόπους. Ένα από τα αιτήματα του επιτρόπου στο οποίο συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα, του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα, ήταν η σύσταση μιας ε, διοντολογική επιτροπής που θα εξέταζε τα θέματα σύγκρουση συμφερόντων πριν και κατά την ανάληψη πριν την ανάληψη των καθηκόντων και μετά το πέρας της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πιστεύω ότι στο μέλλον, όπως πρότεινε και η εκλεγμένη πρόεδρος, θα χρειαστούμε έναν ανεξάρτητο τέτοιο φορέα, μια ανεξάρτητη ε, αρχή ιδεοντολογίας. Και με βάση την προηγούμενη μου πείρα θα έλεγα ότι ε, είναι θα χρειαζόμασταν κάποιον που θα έχει πείρα ή θα πρέπει να στηριχθεί πείρα, στην πείρα ανθρώπων που γνωρίζουν τις διοργανικές σχέσεις και δεν θα είναι χρονοβόρη η διαδικασία ε, έκδοση των αποφάσεων και θα στελεχώνεται αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή από ανθρώπους που φυσικά θα επιτελούν με ανεξαρτησία το έργο τους. Αν έχετε περώτηση πραγματικά θα πρέπει να είναι επιγραμματική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την απάντηση. Όντως, ε, χρειάζονται μέσα για την ανεξαρτησία και σε σχέση με τη διαφάνεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Απαντήσατε εν μέρη, αλλά κάποιες χώρες ε, μπροστά στις κάμερες υιοθετούν προοδευτικές απόψεις και στις ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου ε, λένε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ανάγκη διαφάνειας για όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και επίσης ο δεοντολογικός κώδικας είναι πολύ σημαντικό θέμα και δεν θα πρέπει να γίνονται αδιαφανείς αποφάσεις ε, ιδιαίτερα στα θέματα τα φορολογικά από το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα της διαφάνειας να εξεταστεί σε όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι προφανές και από την σημερινή συζήτηση ότι αυτό το θέμα μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές είναι προσφυλέ σε όλου του επιτρόπου και φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα προσφυλέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα τη διαφάνεια. Θα το διαβιβάσω λοιπόν το μήνυμά σα στο Συμβούλιο και θα προτείνουμε ε, μέτρα για τη συνέχεια. Πάντως, η Φιλανδική Προεδρία πρότεινε διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνεια. και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάτι που θα σας ικανοποιεί. Βέβαια, πολλές χώρες είναι υπέρ της τις ε, θαραλές αυτής τάση της Φιλανδικής Προεδρίας και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω τις συζητήσεις και με την επόμενη Προεδρία για να βρούμε ικανοποιητικές λύσεις για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και στο Συμβούλιο. Επόμενη ερώτηση από, την, από τον κύριο Χαϊσέλ, Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω την ερώτηση στα ε, σλοβακικά, λέει ο κύριος Χάισελ. Ε, Κύριε Σεφτσοβίτς, στη νέα σας ομάδα έχετε ε, νέα εντολή να ε, βλέπετε και να εντοπίζετε τις νέες τεχνολογικές τάσεις. Αυτό θα επηρεάσει και την τεχνολογία μας και την οικονομία μας, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση. Εδώ η Ευρώπη θέλει να είναι ανταγωνιστική, ε, αλλά και πρωτοπόρα εκτός από ανταγωνιστική. Παγκόσμιος ηγέτης. Εσείς είστε τρόποντινά Ε, στην πρώτη γραμμή ε, ε, στη συμμαχία για τις μπαταρίες. Τι λείπει όμως από την Ευρώπη για να είμαστε πραγματικά στην πρώτη θέση. Τι να κάνουμε έτσι ώστε τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα να εξάγονται από την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο. Γιατί να μην σχεδιάζουμε απλώς εμείς τα αυτοκίνητα αλλά και να τα παράγουμε. τι πρέπει να κάνουμε εκεί έτσι ώστε να καλύψουμε τη διαφορά που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρόνια που έχουμε τα δύο-τρία. Ε, απάντηση στα σλοβακικά επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Αυτό που δεν είχαμε εδώ πριν από δύο-τρία χρόνια ήταν η ε, συνειδητοποίηση ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πραγματικά το μέλλον της ε, κινητικότητας. Ε, και αν δεν ε, καταλάβουμε κάτι τέτοιο και δεν ε, είμαστε κυρίαρχοι αυτού του μέλλοντος, δεν θα είμαστε ποτέ σε πρώτη θέση ε, από πλευράς κατασκευής αυτοκινήτων. Σήμερα ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βιομηχανική τέτοια συμμαχία. Έχουμε πάνω από 200 εταιρείες που ενέχονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής του κλάδου αυτού. Ας πούμε, έχουν συγκεκριμένους πόρους, ε, σύγχρονα λογισμικά και τεχνολογίες ε, ε, δυνατότητας αποθήκευσης ενέργειας και στη συνέχεια μεταπόλησης του στα δίκτυα. Οι δικές μας μπαταρίες, αυτές που θα παράγουμε εμείς, θα πρέπει να είναι οι πιο πράσινες, οι πιο οικολογικές για να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται και στη μηχανία ή ακόμα και στα νοικοκυριά. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και μεγάλη. Και τώρα εμείς τι θέλουμε, τα ε, καθαρότερα αυτοκίνητα να κατασκευάζονται πραγματικά στην Ευρώπη. Αυτά θα πρέπει να κωδικοποιηθούν νομοθετικά ε, και ως προς τα πρότυπα και τους κανόνες να είναι συγκεκριμένοι. Εάν θέλουμε να έχουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Ευρώπη, τότε αυτό θα γίνει μόνο με υψηλά πρότυπα που θα μας παρέχουν οι καλύτερες, πιο οικολογικές, πιο πράσινες μπαταρίες οι οποίες θα παράγονται και στην Ευρώπη. Και ταυτόχρονα υπάρχει και το θέμα των επενδύσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί. Οπότε δεν ανησυχώ πάρα πολύ όπως ανησυχούσα παλαιότερα. Ε, συμπροματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή ερώτηση, κύριος Χάισελ. Αυτή η μετάβαση ε, μπορεί να αποδειχθεί επώδυνη. Ρωτώ, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε αυτούς τους φόβους και τις αγωνίες των ανθρώπων που φοβούνται, μήπως χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. Τι θα κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε και από την κοινωνική σκοπιά ε, να υπάρχουν όσο γίνεται ε, λιγότερες επιπτώσεις και ε, να είναι λιγότερο οδυνηρή αυτή για τους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την επερώτησή σας. Εμείς ως ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετύχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Γιατί ε, επιβάλαμε να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης των περιοχών που παράγουν άνθρακα, για παράδειγμα. Και στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα ληφθεί υπόψη η μετάβαση σε αυτές τις περιοχές. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Πριν από δύο-τρία χρόνια ήταν κάτι τέτοιο αδιανόητο. Το ίδιο ισχύει και για τη συμμαχία για τις μπαταρίες. Ε, θα πρέπει να έχουμε ένα πρότυπο για το πώς θα τοποθετηθούμε εκεί και απέναντι σε άλλους τομείς που πρέπει να είναι ε, ισχυρή Ευρώπη. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις περιφέρειες αυτές για το μέλλον, να βγούμε να πούμε από τώρα ότι είναι σωστό και σημαντικό να αλλάξουμε ε, την παραγωγή, ότι χρειαζόμαστε νέες εταιρείες. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και σε κάποιους άλλους κλάδους της βιομηχανίας που υπολείπονται, έχουν μείνει πίσω δύο-τρία βήματα. Χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες και νέες γνώσεις για τους ανθρώπους σε αυτό το κλάδο. Ο κύριος Σέμς Ρώτο από το Κόμμα των Πρασίνων και την Επιτροπή Αναφορών. Mr. Vice President, as an expert on foresight, you already know what ως ε, ειδικό ε, στις προβλέψεις και στον προγραμματισμό θα ξέρετε ήδη τι θέλω να πω. Εφόσον τίποτα δεν μπορεί να σας εκπλήξει θα είστε πολύ χαλαρός. Σας ζηλεύω. Εγώ δεν ξέρω καν τι θα ε, μου συμβεί αύριο. Τι θα γίνει. Α, αυτή η, η αγωνία με τρελαίνει. Τι θα γίνει λοιπόν μέχρι το 2024 σε αυτή τη σαστηθετία σε σχέση με την ε, ανθιγινή σχέση μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και της Κομισιόν. Ε, ε, έχετε, έχετε αρχίσει, μάλλον θα αρχίσετε μία θεραπεία ζευγαριού. Μετά, σε σχέση με την νομοθεσία και με τη θέση σας θα εξασφαλίσετε ότι οι επίτροποι δεν θα έχουν να κάνουν με σύγκρουση συμφερόντων ούτε και με προέδρους που μπορεί να έχουν στενές σχέσεις με διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες και συμβούλους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σέμστροτ για τις ερωτήσεις σας. Όταν ε, μου επιδόθη το χαρτοφυλάκιο για τι προβλέψεις, κάποιοι συνάδελφοι αρχίζαν να με ρωτάνε τα νούμερα του Λότο ε, για την επόμενη κλήρωση. Δυστυχώ δεν έχω τέτοιε ε, μαντικές ε, ικανότητες και οι προβλέψεις που λέμε εμεί δεν αφορούν ε, καμιά κρυστάλλινη μπάλα, αλλά σφαίρα, αλλά να δούμε αν και πω η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πώς θα είναι η Ευρώπη το 2030-40, πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Και έπειτα πιστεύω πως η επιστήμη θα μας δώσει καλές συμβουλές, θα τα καταφέρουμε. Ε, όχι όμως να συνεχίσουμε με τις σημερινές πολιτικές. Εάν βελτιώσουμε λίγο τις προσπάθειές μας, ναι, ε, ε, θα τα καταφέρουμε κάπως καλύτερα. Όμως τι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό το σενάριο να γίνει πραγματικότητα και πώς θα, θα προβούμε στα απαραίτητα βήματα στον οικονομικό τομέα, στην νομοθεσία, στους ρυθμιστικούς τομείς, ώστε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά να κατασκευάσουμε την πράξη ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Αυτό θα πει η πρόβλεψη, προγραμματισμός. Ε, όχι μόνο να παρουσιάσουμε δηλαδή το μέλλον, αλλά να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για, και, με ποιον τρόπο και με ποιες προσπάθειες θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Τώρα, για θεραπεία ζευγαριού δεν χρειάζεται, ε, νομίζω, μεταξύ Επιτροπής ε, και Επιτροπής Αναφορών, γιατί συνήθως ε, τα προβλήματα των ζευγαριών είναι προβλήματα επικοινωνίας. Γι' αυτό σας λέω ότι θα είμαι όσο θέλετε εκεί να απαντώ και στις ερωτήσεις σας και για το θέμα του δικαιώματος των πολιτών. Έχουμε αποδείξει ότι αν ε, πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων, είστε σκληροί και δεν θα διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τις αρμοδιότητές σας και αυτό δεν με φοβίζει καθόλου. Η αποστολή σα λέει, η εντολή σα λέει πω είστε υπεύθυνο για το διάλογο ανάμεσα στου ανθρώπου και την Κομισιόν. Εσεί όμω αυτό που σκοπεύετε να κάνετε είναι ένα μονόλογο. Αν θέλετε ο κόσμο να ενδιαφέρεται για το τι κάνει η Ευρώπη, θα πρέπει να του δώσετε το λόγο. Θα πρέπει να του δώσετε μάλλον δυνατότητα να πούν τη γνώμη του και εκείνοι. Ε, υπάρχει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο που θα μπορούσε να απελευθερωθεί και οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν περισσότερα από εσά, που ε, είναι πιο δημιουργικοί από εσά και που θα έκαναν τη δουλειά σα και για λιγότερα λεφτά. Τώρα, αν ξαναδούμε την κρυστάλλινη σφαίρα, τι κάνατε ακριβώς για να δώσετε σε αυτόν τον κόσμο όλο περισσότερη εξουσία. Νομίζω πως ε, έχουμε καταφέρει πολλά. Αν έπρεπε να δω τη δική μου απόδοση, να αξιολογήσω τη δική μου απόδοση των τελευταίων 10 χρόνων, ήμουν ένας από τους πιο τακτικούς συνομιλητές με τους πολίτες ε, στον διάλογο με τους πολίτες και μάλλον ε, επισκέφθηκα τα περισσότερα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και περιφερειακά συμβούλια. Όχι επειδή είμαι καλός, αλλά επειδή έχω ε, μεγαλύτερη θητεία και ήταν το καθήκον μου. Και τώρα η πρόεδρο θέλει να κάνουμε όλοι μα το ίδιο, να επισκεφτόμαστε τα κράτη-μέλη μέσα στο πρώτο ήμιση τη εντολή, όλα. Και βεβαίω δεν θα μιλήσουμε με του ε, υπουργού ή μόνο του βουλευτέ. Θέλουμε να συνομιλήσουμε με του πολίτε. και θα ήθελα συγκεκριμένε προτάσει για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Γιατί διαβουλευόμαστε με τον κόσμο μέχρι τη πλατφόρμα Have Your Say. Πε και εσύ τη γνώμη σου. Αλλά δεν είναι ιδανικό, το ξέρω. Προσπαθούμε να σκεφτούμε διάφορους τρόπους να χρησιμοποιήσουμε το Facebook σε πλατφόρμα για να μιλήσουμε με τους νέους. Ε, ε, ε, πώς μπορούμε να, δηλαδή, να, να αγγίξουμε τους νέους, ε, να είμαστε δημιουργικοί. Οι νέοι θα μας πούνε πώς θα κάνουμε καλύτερα αυτή την επαφή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να μάθουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρνς από το Ρινιού μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις ε, μικτές αρμοδιότητες, κοινές αρμοδιότητες, ε, ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο λόγο εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ αποδοτική. Ενώ οι συνθήκες μιλούν για την επιτακτική ανάγκη του συντονισμού που κατοχυρώνεται στην συνθήκη της Λισαβόνας. Για παράδειγμα, θέματα δημόσιων ενισχύσεων ε, για την ανάπτυξη, δημόσια αναπτυξιακής βοήθειας. Εδώ και μισό αιώνα έχουμε κάνει αυτή την υπόσχεση και την ε, παραλαμβάνουμε μονίμως στις ε, διεθνείς διασκέψεις και στο Συμβούλιο ε, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για το 0,7% σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά μόνο τέσσερα κράτη έχουν τηρήσει την υπόσχεσή τους. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Θα αρκεστείτε σε απλή αναφορά της ε, έλλειψης αρμοδιότητας ή θα ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν περισσότερο τις ευθύνες τους. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και σας ευχαριστώ για το απτό παράδειγμα που δώσατε. Έχετε δίκιο. Πολύ συχνά οι φιλοδοξίες που ακούγονται στη συνεδρίαση και στις συνεντεύξεις τύπου είναι πολύ ψηλότερες από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και την τελική έκβαση υπάρχει το θέμα της πολιτικής πραγματικότητας. Και σίγουρα στην αμοιβαία συνεργασία μας θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας και να τις αναβαθμίσουμε. Και εκεί θα παίξει ρόλο και η πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό όμως που βλέπω κυρίως στα κράτη-μέλη είναι μεγαλύτερη πίεση των ομοτήμων. Μεγαλύτερη απέτηση για να τηρηθούν τα υποσχέσεις και οι δεσμεύσει, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τους στόχους τους. Πολύ συχνά όταν μιλούμε για τα προβλήματα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, μερικές φορές αυτά οφείλονται σε κακοδιαχείριση, έλλειψη διοικητικής ικανότητας ή μη σωστή αντίληψη του τι πρέπει να γίνει αλλά θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και να τα εξοπλίσουμε καλύτερα για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις τους. Και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι αυτό της αναπτυξιακής βοήθειας που αναφέρατε. Και αυτό θα είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η επόμενη Επιτροπή. Και σίγουρα η συνάδελφος Ουρπιλάινεν θα είναι αρμόδια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα, θα συνεργαστεί, φαντάζομαι, πολύ στενά και εκείνη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεπεράσουμε το κενό που ήδη υπάρχει, το χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων, των υποσχέσεων των κρατών μελών για την αναπτυξιακή βοήθεια και των αποτελεσμάτων. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα από το Ταμείο του Γιούγκερ, ώστε οι εξωτερικές μας επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές και θα μπορούσαν να αποφέρουν περίπου 40 δισεκατομμύρια για σωστά σχέδια στην Αφρική, που είναι αυτό που χρειάζεται η Αφρική, καλά προγράμματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί καλύτερα να τα χρηματοδοτήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι όλα τα προσπαθήσαμε. Έκκληση ε, στη φιλότιμο, στη λογική, στην τήρηση των υποσχέσεων, αλλά όλα αναβάγησαν. Ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως ε, βρήκε με μια συνθήκη τα μέσα να φέρει τους υπουργούς προϋπολογισμών στην Αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λογοδοτήσουν για αυτά που έκαναν ή για αυτά που αμέλησαν να κάνουν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για ένα μηχανισμό και να φέρουμε και τους μηχανισμούς ανάπτυξης στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λογοδοτούν για τις παραλήψεις τους. Και νομίζω ότι το σύστημα είναι προβληματικό, γιατί το σύστημα είναι αναποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Ίσως όντως ήταν χρήσιμο να έχουμε στενότερες επαφές μεταξύ των αρμόδιων ε, υπουργών για την αναπτυξιακή βοήθεια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλύτερη, πιο στενή σχέση. Έτσι θα ε, αυξηθεί η δημοκρατική πίεση και η πίεση ομοτήμων των χωρών, ενώ που ανέλαβαν υποσχέσεις και δεσμεύσεις, αλλά δεν τις στήρισαν. Επίσης, έτσι θα δημιουργηθεί και η μεγαλύτερη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη και να βρει άλλους τρόπους για να τα ενθαρρύνει να τηρήσουν την υποστήριξη που υποσχέθηκαν και όχι μόνο τα δημοσιονομικά μέσα. Μόχλευση, χρήση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επίσης ένα τμήμα που θα μπορούσε να περάσει στο Ταμείο για το Κλίμα, να βρεθούν χρήματα για να ε, χρηματοδοτηθούν προγράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες για να έχουν αποτελέσματα πιο άμεσα προς όφελος των πολιτών τους. Και η τελευταία ερώτηση για το απόγευμα θα υποβληθεί από τον κύριο Ρανζέλ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. <clears throat> Ε, κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά. Και θα ήθελα μέχρι την τελευταία ερώτηση να κρατήσω το θέμα του ελέγχου ε, απαντήσατε και γραπτός και προφορικά σήμερα και ακούγοντας όλα αυτά κανείς τι είναι να πιστεύει ότι θα είστε μάλλον ε, επίτροπος διοργανικών σχέσεων και λιγότερο για τις προβλέψεις. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη φιλοδοξία γιατί αλλιώς υποτίθεται ότι θα είστε αντιπρόεδρος για τις διοργανικές ε, σχέσεις και το status quo αντί για τις προβλέψεις. Διαπραγματευτήκαμε μαζί το 2010 τη διοργανική συμφωνία και είπατε ότι καλό θα ήταν συμπεριλαμβάνει και το Συμβούλιο. Ποια είναι όμως τα συγκεκριμένα βήματα που προτίθεστε να αναλάβετε και επί της ουσίας τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει. Το Συμβούλιο όλο και περισσότερο ε, τι είναι να γίνει μια γερουσία. Το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να έχει ε, περισσότερη πρόσβαση στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή σωστή πρόσβαση στα έγγραφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρανζέλ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή θα προσπαθήσω να αυξήσω τη φιλοδοξία μου για το μέλλον στις επιδόσεις μου. Και σας ευχαριστώ για την τεράστια βοήθεια, υποστήριξη και τις συμβουλές που έλαβα από εσά καθ' όλη τη δύσκολη περίοδο των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Και θυμάμαι πάρα πολύ πως και οι δυο μας είχαμε απευθύνει έκκληση στο Συμβούλιο να συνεργαστεί σε αυτή τη συμφωνία. Και θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε μια πιο ισόρροπη ε, ε, διαδικασία για το πώς ε, προσαρμόζουμε στη συνδίκη της Λισαβόνα στην καθημερινή δουλειά και των τριών θεσμικών οργάνων. Εκείνη την εποχή κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, κυρίως επειδή υπήρχαν διάφορες νομικές έτσι, ανησυχίες και αντιρρήσεις από πλευρά Συμβουλίου. Από τότε όμως έχει περάσει πολύς χρόνος και έχουν μεσολαβήσει πολλά. Κατευθύσαμε να έχουμε μια τριμερή συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Και χαίρομαι επίσης που κάθε χρόνο ε, βγάζαμε κοινή δήλωση για ανακοίνωση για τα στρατηγικά βήματα για το ε, επόμενο έτος κάθε φορά που έπρεπε να εστιάσουμε. Παρόλο που είναι σχετικά νέο το σύστημα, νομίζω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Προτείνω λοιπόν το εξής και προς το Συμβούλιο και προς εσάς. Να δούμε πώς εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία πλαίσιο. Μπορούμε να ε, συμπεράνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει αυτό τη σύνδικη της Λισαβόνας, αλλιώς θα είχαν προσφύγει στο δικαστήριο. Και πώς ε, μπορούμε να πείσουμε το Συμβούλιο ότι αφού έχουμε τόσο καλές σχέσεις μεταξύ μας, καλό θα ήταν και θα ήταν και πιο ευεργετικό για όλους και πιο αποδοτικό για να έχουμε καλύτερες ε, διοργανικές σχέσεις. Με χαρά ε, σηκώνω το γάντι και θα μιλήσω στις προεδρίες. Και αφού όταν με εγκρίνετε ελπίζω θα έχω την ευκαιρία να συμμετέχω στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Χρειαζόμαστε ε, συνεργασία και για τις στρατηγικές συζητήσεις και για τις ε, ε, πολιετίες που θα πρέπει να κάνουμε μαζί. Συμπροματική ερώτηση από τον κύριο Ρανζέλ. Μιλήσατε για την ευθύνη σας και για τη σχέση μας Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν μιλούν εξ ονόματος άλλων επιτρόπων, όχι πάντοτε, αλλά κυρίως κάνουν ε, την εισαγωγική τους τοποθέτηση διαβάζοντας ένα κείμενο έτοιμο. Αλλά και στο τέλος πάλι ε, συμπερασματικά καταλήγουν διαβάζοντας ένα κείμενο που φαίνεται να έχει συνταχθεί πριν την έναρξη της συζήτησης. Άρα λοιπόν, για τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεισφορά στη, ε, συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι ε, κάτι που αρμόζει. Και αν όχι, πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. I have to admit that you are right. Ομολογώ, είμαι υποχρεωμένος ότι έχετε δίκιο. Ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα θέμα κάποιου συναδέλφου, τελευταία στιγμή ε, που τον αναλαμβάνουμε, ε, είναι γεγονό ότι μας δίνουν κάποια εισαγωγικά σχόλια και κάποια καταληκτικά σχόλια. Ε, και βέβαια αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το χρόνο που έχει ο Επίτροπος για να μάθει ένα θέμα που του είναι άγνωστο, καινούριο. Η είναι. Εσείς τι ζητάτε, σεβασμό προς τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι σας ακούμε. Γιατί κάνετε προτάσεις τις οποίες σημειώνουμε, ε, επεξεργαζόμαστε και απαντούμε ε, στις συγκεκριμένες σας ε, υποδείξεις ή σχόλια στα καταληκτικά δικά μας. Γιατί αυτό που θέλετε είναι να μεταφέρουμε στα θεσμικά όργανα τις προτάσεις σας και να τα επεξεργαζόμαστε. Αυτό σίγουρα χωράει βελτίωση από πλευράς μας και αν μου επιτρέπετε να σας προτείνω, θα μας βοηθούσε περισσότερο ε, αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιος θα πάει στην Ολομέλεια. Αυτό είναι στα χέρια σας και αν μπορείτε εσείς να το διευκολύνετε, θα μας διευκόλυνε και εμάς πάρα πολύ. Thank you very much for your question. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και όλες τις ερωτήσεις που ήταν ε, εξαιρετικές. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σεφτσοβίτς για πέντε λεπτά για τα καταληκτικά του σχόλια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μάθω από την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Ρανζέλ. Θα αντιδράσω ενθερμό στα, στη σημερινή συζήτηση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι καθίσατε σαφές πόσο σημαντική είναι η αγαστή σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Πολλές από τις προτάσεις σας ε, σήμερα ε, είναι πηγή έμπνευση για τη μελλοντική μου εργασία. Πολύ με ενθαρρύνει η στάση σας να φέρετε νέες μεθόδους, ε, νέες προσεγγίσεις για το πώς νομοθετούμε, πώς πώς συνεργαζόμαστε και πώς ε, ε, προσφέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στους συμπολίτε μας. πρέπει νομίζω να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε περισσότερο γιατί είμαι απόλυτα βέβαιος πως τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν το πεπρωμένο της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα σηματοδοτήσουν τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, όχι μόνο τον κόσμο το 2030, αλλά για ολόκληρο τον υπόλοιπο αιώνα. Πιστεύω πως όλοι μας επιθυμούμε η Ευρώπη να είναι καθαρότερη, πρασινότερη, πιο αποδετική, πιο κοντά στους πολίτες και να παίζει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο ε, στις, ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Όταν κανείς ταξιδεύει εκτός Ευρώπης, αυτό που ακούει είναι όχι μόνο κομπλιμέντα για το πόσο καλά συνεργάζονται μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ε, και εκκλήσεις ώστε εμείς οι Ευρωπαίοι να, είμαστε, ε, να έχουμε περισσότερη επιρροή ε, από ό,τι μέχρι σήμερα. Γιατί σέβεστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, σέβεστε τη φύση, σέβεστε το διεθνές δίκαιο, προσπαθείτε να είστε όσο γίνεται πιο υπεύθυνοι ε, προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, επειδή είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε και να συμβάλλουμε. Και χάρη σε αυτά μας τα χαρακτηριστικά η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς στη γη. Είναι λοιπόν στρατηγική η θέση μας, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να ανταποκρινόμαστε στους πολίτες μας και πιστεύω πως εάν έχω την, την ε, ψήφο σας θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας για όλους αυτούς τους τομείς ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτή την πολύ φιλόδοξη ατζέντα στους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές σα ερωτήσεις και για να ευχαριστήσω επίσης τους δύο προέδρους των Επιτροπών Επιτροπών για την αυστηρή Προεδρία, αλλά πολύ ευγενική Προεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. On behalf of the Εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, υποψήφιο αντιπρόεδρο για τη διεξοδική απάντηση ερωτήσεις που έδωσε και την προσοχή με την οποία άκουσε τις ερωτήσεις. Πραγματικά φάνηκε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και σίγουρα η πολιτική one in, one out θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της επόμενης Επιτροπής. Έχετε το χαρτοφυλάκιο το, της πρόβλεψης, της διορατικότητας. Όντως, χρειαζόμαστε τεκμηριωμένη νομοθεσία. Νομοθεσία που θα στηρίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και επίση να χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία αποτελεσματικά αλλά και με δεντολογικό τρόπο, με ηθικό τρόπο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν για τις εμπεριστατωμένες και διεξοδικές μας σας απαντήσεις και ευχαριστώ που λάβατε μέρος στην απόψηνή μας δημόσια κρόαση. Και εγώ θέλω να προσθέσω τις δικές μου ευχαριστήσεις, τις ευχαριστήσεις Επιτρόπου Γιούρη για τη διαθεσιμότητά σας, αλλά και επειδή επιδείξατε μεγάλο ενδιαφέρον απέναντι στο Ευρωκοινοβούλιο. Το έχετε δείξει στο παρελθόν. Ξέρω πόσο έχετε κάνει όταν ήμουν και εγώ, ήμασταν μαζί οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και στην προηγούμενη θητεία ανέκαθεν είχατε πολύ ψηλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς ε, δεν το έπραξαν αυτό, αυτό οι, όλοι οι προηγούμενοι Επίτροποι. Κάποιες φορές μάλιστα ήταν και υποτιμητικοί απέναντι στο Κοινοβούλιο, σαν να ήταν θυσία δηλαδή να έρθουν εδώ και να συνομιλήσουν με το Ευρωκοινοβούλιο έκαναν. Εσείς απαντήσατε πολύ συγκεκριμένα στις ερωτήσεις μας, ε, δεσμευτήκατε να έρθετε στις επιτροπές και να συζητήσετε μαζί μας κάθε φορά που θα προσκληθείτε. Αλλά εσείς δεν είστε ένας οποιοδήποτε επίτροπος, είστε αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Και γι' αυτό και σας ζητούμε βεβαίως να ασκήσετε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ε, ε, το έργο σας ως συνομιλητή της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, αλλά να κυρίως να εξηγήσετε σε όλους τους επιτρόπους και κυρίως τους νέους επιτρόπους πόσο σημαντική είναι η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Καθήκον μας είναι να ελέγχουμε την εργασία σας ακριβώς έτσι ώστε να δίνουμε καλύτερες απαντήσεις στους πολίτες. Γι' αυτό και σας ζητώ και επειδή σας γνωρίζω εδώ και τόσα χρόνια να ασκήσετε το ρόλο του Αντιπροέδρου και προς του συναδέλφου σα ώστε και εκείνοι να έχουν αυτή την ευαισθησία που εσείς έχετε δείξει τα τελευταία χρόνια, ότι οι σχέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικές και συχνά είναι σημαντικό να υποστηρίζετε την Επιτροπή στα brand fair που έχουμε με το Συμβούλιο. Συχνά το Συμβούλιο προστατεύει εθνικά συμφέροντα και δεν καταφέρνει να ενεργήσει με ευρωπαϊκή υπευθυνότητα. Εμείς στο, στην, εποχή της παγκοσμιοποίησης θα είμαστε αδύναμοι αν δεν είμαστε ενωμένοι. Προφανώς και υπάρχουν εθνικές ευαισθησίες, αλλά η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο που εκπροσωπούν ε, τα πιο κοινοτικά θεσμικά όργανα, ας πούμε, ε, να πείσουμε και το Συμβούλιο, ας πούμε, το μπλοκάρισμα του Δουβρίνου που εμείς θέλαμε, η Κομισιόν ήθελε, αλλά τα κράτη-μέλη το μπλόκαραν, ας πούμε. Κοινέ ενέργειες και δράσεις θα πρέπει να μας επιτρέψουν να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη και πιο ικανή να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών. Βασιζόμαστε σε εσά και στο έργο σα και όπω έχετε δείξει και στο παρελθόν, είμαστε βέβαιοι ότι θα το κάνετε και στη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Σα ευχαριστούμε που απαντήσατε λοιπόν στι ερωτήσει μα. Ανακοινώσω πω θα γίνει κοινή συνεδρία των συντονιστών για την αξιολόγηση τη ακρόαση που θα ξεκινήσει στις 6 ε, και μισή και κλεισμένων των θυρών λοιπόν θα συνεδριάσουν οι συντονιστές ε, των Επιτροπών Τζούρι και Αύκο και Οι συνεδεμένες επιτροπές θα συνεδριάσουν με τους συντονιστές τους ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ με όλους και λέει, δουλειά.